Ach, 96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

Good If you could uh, make your way Καλησπέρα σας. Αν μπορείτε να καθίσετε. Συνειδητοποιώ βέβαια ότι είστε όλοι πολύ ενθουσιώδεις που συναντιέστε με άτομα των κοινοβουλίων.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 time she comes here. Okay. Right. Um, sorry for this, this slight. We, we, are, we are running concurrent. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Λειτουργούμε ταυτόχρονα με το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και μας ενημερώνουν διαρκώς για το πόσοι πότε θα τελειάσει γιατί η κυρία Σαλγάδος, πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα. Θα προσπαθήσει όμως να είναι μαζί μας πολύ σύντομα. Καλώς ορίσατε στην ετήσια συνέλευσή μας ε, με τους αντιπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται σήμερα και με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και με μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα είναι μια καλή χρονική στιγμή για να συζητήσουμε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης της κρίσης, ανεργίας κτλ. Αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και είναι καλό να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωσή της για την στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέχρι το 2020. Οπότε θα θέλαμε σήμερα να σας ενημερώσουμε και για τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας όπου θα γίνει η παρουσίαση αλλά και γενικότερα για τις συνιστώσεις της στρατηγικής για το 2020. Σήμερα θα συζητήσουμε το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενώ αύριο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αλλά με μια πιο παγκόσμια και συνολική προοπτική. Θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω και τον συμπρόεδρό μου, τον Τζόρντι Βιλατζοάνα, από την Ισπανική Γεωρουσία, που είναι, όπου είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικής Πολιτικής. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Να πω όμως ότι σήμερα θα ακούσουμε την κυρία Ελένα Σαλγάδο όταν θα μπορέσει να έρθει τον κύριο Όλι Ρεν, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα, τον κύριο Γιούργεν Στάρκ, μέλο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τέλος ε, τον κύριο Ζαν Πιζάνη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μπρούγκελ. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο, τον κύριο Τζόρντι Βίλα για να σας πει και αυτός μερικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. να ευχαριστήσω επίση και όλου όσοι κατέβαλαν προσπάθεια προκειμένου να ξεβρεθούν σήμερα ανάμεσά μα. Η συνάντηση αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια μια περίοδου όπου το δείχνει, τα πράγματα δείχνουν ότι το 2010 θα είναι ε, το έτο έναρξη τη ανάκαμψη. Αλλά σύμφωνα με τα όσα λένε οι εμπειρογνώμονε, αυτή η ανάκαμψη θα είναι αργή, εύθραυστη και θα είναι μια ανάκαμψη άνηση. Θα είναι αργή διότι η μηχανή της οικονομίας μας δεν θα έχει την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου που της λείπει αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και μια και μια μείωση των δημοσίων δαπανών. Θα έχουν υπάρξουν όμως και άλλες τροχοπέδες που όπως σε ό,τι αφορά την Ισπανία θα είναι το χρέος των επιχειρήσεων, το χρέος των οικογενειών αλλά επίσης και το χρέη του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχει περιορίσει την δανειοδότηση. Όλα αυτά λοιπόν περιορίζουν τις δραστηριότητες και ως εκ τούτου έχουμε και ως συνέπεια τη μείωση των εξαγωγών μας. Εκτιθέμεθα λοιπόν σε ε, συνεχείς ε, επιρροές, πολλές από αυτές έρχονται από το εξωτερικό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα ποσοστά ανάπτυξης ε, κάποιων κρατών αλλά επίση, ε, εμεί στην Ισπανία δεν ξεχνάμε ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα. Είπα ότι θα είναι άνηση αυτή η ανάπτυξη, διότι δεν θα πετύχουμε τον αυτό ρυθμό σε όλα τα κράτη, ούτε ακόμα και στο εσωτερικό κάθε χώρα, διότι κάθε τομέα θα επηρεαστεί διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ Πρόεδρε θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό που συναντιόμαστε και να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις όλων, να ακούσουμε λοιπόν ποια θα είναι η στρατηγική την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε για να πετύχουμε μια ανάπτυξη πολύ πιο σταθερή, κάτι το οποίο θα αυξήσει και την απασχόληση. Όπως ξέρετε στην χώρα μου έχουμε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτήν την ανάπτυξη προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ενέργεια. Ελπίζω να είμαστε αποτελεσματικοί στη σημερινή μας συνάντηση ε, και στην αυριανή επίση ε, και να προσπαθήσουμε να ξέρουμε λύσεις για την έξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους αν να πούνε κάποια πράγματα μέχρι να φτάσει η κυρία Σαλγάδο. Είναι η δεύτερη ομιλήτρια σύμφωνα με το πρόγραμμά μας και παρακαλώ αν κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο παρακαλώ και το πρόγραμμα είναι να έχουμε τρεις ομιλητές αρχικά και μετά θα ακούσουμε τα μέλη τόσο των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Παρακαλώ πολύ αν ε, θέλετε να λάβετε το λόγο μπορείτε να σηκώνετε το χέρι σας και ο Αντόλφου εδώ θα σημειώνει τα ονόματά σας και από καιρούς καιρών ε, θα ελέγχω και τον κατάλογο των ε, αγοριτών. Και μετά θα επανέλθουμε στους ομιλητές που προβλέπονται από το πρόγραμμα και θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο της συνεδριάσεως. Α, έχετε ζητήσει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Δεν άκουγα την ε, διερμηνία στα Μαλτέζικα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή είναι δικό μου. Ναι, ελέγχουμε, παρατηρεί η Πρόεδρος, αλλά υπάρχει διερμηνία προς και από τα Μαλτέζικα νομίζω. Α, συγγνώμη, λάθος έκανα. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει σήμερα διερμηνία από και προς τα Μαλτέζικα. Ελπίζω να μην σας δημιουργεί ιδιαίτερη, ιδιαίτερο πρόβλημα. Μα, με απασχολούσε το ζήτημα των ε, προσκεκλημένων μας ε, Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις γλώσσες. Μερικές φορές είναι και θέμα αριθμού διερμηνευτικών θαλαμίσκων που δεν επαρκούν. Παρακαλώ. Ο κύριος Κάμπα. είναι Υφυπουργό ε, Οικονομικών ε, στην Ισπανία. Αν θέλετε παρακολουθείτε πείτε μερικά λόγια μέχρι να φτάσει η ε, Υπουργό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την Υπουργό. Α, αυτή τη στιγμή εισέρχεται στην αίθουσα έρχεται από ένα γεύμα που είχαμε με τους υπουργούς και τον πρόεδρο του Συμβουλίου για το ίδιο αυτό ζήτημα, για την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020. Okay, now, now, uh, Εντάξει, τώρα ολοκληρώθηκε η σύνθεση. Ερχόσαστε απευθεία από το ΕΚΟΦΗΝ και σας καλωσορίζω, κυρία Σαλγάδο. Μπορείτε αν θέλετε να περάσετε στην ε, ομιλία σας, εκτός αν θέλετε να ξελαχανιάστε. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και θα μιλήσω την Ισπανική. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα η συμμετοχή μου σε αυτήν την έκτη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχηθώ καλό απόγευμα και βλέπω ότι και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια συμμετέχουν στην σημερινή μας συνάντηση και νομίζω πως αυτό δείχνει το πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει και που θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Να έχουμε λοιπόν εκπροσώπους από όλες τις πλευρές και από όλα τα κοινοβούλια. Η κρίση λοιπόν την οποία γνωρίζουμε κατέδειξε την αναγκαιότητα να βελτιωθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε το εθνικό συμφέρον με το ευρωπαϊκό. Αυτά τα δύο συμφέροντα λοιπόν θα πρέπει να συμπέσουν και αυτό γίνεται μέσα από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευκαιρίες όπως σημερινή μπορούν να συμβάλλουν προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα. Επιπλέον αυτή διακοινοβουλευτική συνάντηση, η οποία συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια, συνεισφέρει σημαντικά στον ενισχυμένο ρόλο που η συνθήκη τη Λισαβόνα αναθέτει τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αναζητώντα όλο και περισσότερο μεγαλύτερη διαφάνεια και μια μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο λοιπόν της μετά την κρίση περίοδο υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απαιτούν ε, ιδιαίτερη προσοχή. προσοχή. έχουμε το σχέδιο για μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση με ορίζοντα δεκαετή το 2020. Ε, Ξάλλου εξυγχρονίζουμε την ε, το ε, γεωμετρία της Ένωσης για να αποφύγουμε στο κρίση όπως αυτή που διανύουμε να επανελειφθεί στο μέλλον. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σήμερα στο πρώτο αυτά τα ζητήματα. Η ευρωπαϊκή στρατηγική μέσω μακροπρόθεσμη ε, είναι ένα από τα θέματα τα πλέον σημαντικά της ευρωπαϊκής ατζέντα και ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέμα, ζητήματα για την Ισπανική Προεδρία. Αυτή η γραμμή δράση λοιπόν αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία στην στρατηγική εξόδο από την κρίση. Τώρα ήδη γνωρίζουμε και έχουμε όλοι αποδεχτεί πως η στρατηγική εξόδο από την κρίση δεν θα πρέπει να ε, επηρεάσει μόνο τα προβλητικά συστήματα ή τα χρηματοπιστωτικά, αλλά η έξοδος από την κρίση θα πρέπει να συμπεριλάβει και στοιχεία τα οποία θα είναι ικανά να οδηγήσουν τις οικονομίες μας σε μια ανάπτυξη πιο ισχυρή, πιο ισόρροπη, πιο βιώσιμη, πιο αηφόρο και δημιουργώντας ε, ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Αυτή λοιπόν θα είναι με καλύτερες εγγύσεις ώστε διαδικασίες που προωθούμε για τη στρατηγική εξόδου αφενός και φορολογική ε, ενοποίηση να είναι το διαρκές Τώρα η επασχόληση για το 2020 μας ε, οδηγεί στο να συντονίσουμε τις πολιτικές μας για να αποφύγουμε κρίσεις όπως αυτή την οποία βιώσαμε. Οι απαιτήσει στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σίγουρα είναι απαραίτητο, αλλά όχι μόνο μεταξύ χωρών, αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τις προτεραιότητες στο πλαίσιο των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και επίσης ε, να δούμε ποιο είναι το σύστημα διακυβέρνησης ε, που θέλουμε να αποκτήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις των προσεχών Η Ισπανική Προεδρία εργάζεται εντατικά σε συνεργασία με την Κομισιόν αλλά και με τη νέα μόνιμη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θεσμικές ε, ανταλλαγές αλλαγές συγγνώμη, μείωσαν σημαντικά το χρονική διάρκεια για την συντονισμό. Φυσικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν, ε, μια συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου εξαμήνου. Ήδη δουλεύουμε προκειμένου να συμφωνήσουμε επί των ουσιοδεστέρων ζητημάτων στο Συμβούλιο το Μάρτιο και τον Ιούνιο να μπορέσουμε να λάβουμε τις επόμενες αποφάσεις. Το Συμβούλιο του Μαρτίου θα αντιδράσει στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ε, μια συμφωνία για την νέα οικονομική στρατηγική και το ποιο θα πρέπει να είναι το γενικότερο σχέδιο διακυβέρνησης. <clears throat> Επειδή ο χρόνος πιέζει, ε, μιλάω για το χρόνο ανάμεσα στην ανακοίνωση Κομισιόν και το Συμβούλιο του Μαρτίου. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας να μπορέσουν να ε, εγκρίνουν κάποια συμπεράσματα στο ΕΚΟΦΗΝ που διεξάγεται σήμερα. Ε, στο Συμβούλιο θα έχουμε ανταλλαγές απόψεων σχετικά με ζητήματα αρμοδιοτήτων, θέματα τα οποία θα προωθηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω έξω ονόματος ως Πρόεδρος του ΑΦΗΝ γνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνουν μέσα, αυτή την και ε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Η κρίση κατέδειξε την ε, σημασία μιας συντονισμένης και κοινή δράσης και η προβολή όλης της στρατηγικής και η ανακοίνωση αυτής της στρατηγικής προς τους πολίτες αναφίβολα θα αποτελέσουν δύο σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της όλης της διαδικασίας. Απαιτείται να ενισχύσουμε με τον συντονισμό, να βελτιώσουμε τις συνέργειες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να υπάρξει κοινή δράση συντονισμένη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η στρατηγική λοιπόν θα δώσει προτεραιότητα στις, ε, στους τομείς που απαιτούνται προκειμένου να βοηθηθούν για την δημιουργία θέσεων εργασία. Προσπαθούμε λοιπόν να ξέρουμε μια στρατηγική πιο απλή αλλά πιο εστιασμένη. Ελπίζω να επιτευχθεί συνένεση σε ό,τι φορά την κινητοποίηση όλων των μέσων για την επίτευξη των στόχων συμπεριβλημένων και των χρηματοπιστωτικών. Επιλέξαμε μια σειρά προτεραιοτήτων και αναζητήσαμε μάλλον και προσπαθήσαμε να βρούμε τους απαραίτητους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτό με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να προδικάσει ποια θα είναι η συζήτηση για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές είναι πιθανόν να υπάρξει συνένεση σχετικά με τις προτεραιότητες ε, δράσεις για τα προσεχή έτη τα οποία, τις οποίες έχει εντοπίσει η Κομισιόν προτεραιότητες που θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ και που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με αυτές που παρουσίασε η Ισπανική Προεδρία στις προηγούμενες συζητήσεις. Ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικό και αηφορία. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, θεμελιώδη θα έλεγα, για την πρόθεση της απασχόλησης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα ώστε να προσεγγίσουμε θέσεις ε, που αφορούν τους ποσοτικούς στόχους, ε, στους οποίους θα εντοπίσει αυτή η νέα στρατηγική θεωρούμε συνειδητό σημαντικό από πλευρά Υπουργών Οικονομικών και Εθνική Οικονομία ε, όλοι αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι, όχι μόνο να ε, είναι δικαιολογημένη, αλλά να είναι ρεαλιστική και φιλόδοξη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνέπεια και συνεκτικότητα ανάμεσα σε αυτούς τους κοινωτικούς στόχους και τους ε, εθνικούς στόχους. Οι στόχοι αυτή που ξέρουμε ότι είναι σημαντική, θα μπορέσουν στην ευκαιρία αυτή να εκπληρωθούν στο σύνολό τους. Αλλά η προσπάθεια συντονισμού θα πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο του νέου συστήματος διακυβέρνησης. Υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάτι το οποίο θα απαιτήσει μια καλύτερη χρήση των μέσων που μας ε, παρέχει η συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να, πιο, να εργαστούμε πιο υπεύθυνα, ειδικά οι χώρες και το Συμβούλιο ε, ε, υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στις ε, δημοσιονομικές πτυχές και την πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις ε, πτυχές της μικρο και της μακροοικονομικές των οικονομιών μας. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει συνένεση σε ό,τι φορά την επιτήρηση των χωρών. Μια συνένεση για θέματα εποπτείας και επιτήρησης Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να επηρεάσουν την φορολογική ε, εποπτεία η οποία θα πρέπει να υπάρχει στο πλαίσιο της, ε, του Συμφώνου Ανάπτυξης ε, και Σταθερότητας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των μακροοικονομικών ανισοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών και να υπάρξει μια εποπτεία πολύ πιο στενή των μεταρρυθμίσεων που έχουν άμεση επιπτώσει στην οικονομική ανάπτυξη. Τονίζω η ιδέα αυτής της ε, εποπτείας ε, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αποδυναμώσει την ε, συνθήκη. Αλλά θα πρέπει να εξετάσει ζητήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής και ιδιαίτερων ελέγχων. Θεωρούμε ότι το να επεκτείνουμε την φορολογική εποπτεία σε άλλους τομείς είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα οριζόντια θέματα θα θεωρώ ότι μπορούν να μας βοηθήσουν στην επίλυση των ε, προβλημάτων. Για να γίνει όμως αυτός ο έλεγχος, αυτή η υποπτία, θα πρέπει να εξετάσουν τα συστήματα πληροφόρηση και αξιολόγηση τα οποία χρησιμοποιήσαμε στο πλαίσιο του ΕΚΟΦΗΝ. Χρειάζεται επίσης να σκεφτούμε το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων μας για να έχουμε μεγαλύτερες επιπτώσεις επί των εθνικών αποφάσεων. Επίσης θα πρέπει να το βλέπουμε ένα νέο σχήμα υπευθυνότητας ε, με καλύτερη ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με πιο ξεκάθαρη ε, ξεκάθαρη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι μόνο το ECOFIN ή το Eurogroup το οποίο ασχοληθούν με αυτήν την ε, στενή εποπτεία. Οι διάφορες, ε, τα διάφορα μέρη του Συμβουλίου θα πρέπει να ασχοληθούν με το θεματικό ζήτημα και τον θεματικό έλεγχο. Θα πρέπει να καθορίσουν λοιπόν μηχανισμούς αφής για να διασφαλίσουμε την συνέπεια ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις της ε, εποπτείας. Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μέσων που μας προσφέρει η συνθήκη. Η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει νέα μέσα για να ενισχυθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις χώρες ευρώ, αλλά και τον συντονισμό ανάμεσα στο σύνολο των κρατών που ε, αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χάσουμε Χρειάζεται επίσης να κάνουμε μια καλύτερη χρήση ενός ουσιώδους μέσου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, όπως είναι η γενική προσανατολισμή της οικονομικής πολιτικής. Θα φροντίσουμε να αποκτήσουμε ε, κάποιες συστάσεις ε, χρήσιμες και διάφανες ε, και με κατάλληλη πρικοδότηση. Η νέα στρατηγική φυσικά θα πρέπει να βελτιώσει την επικοινωνία και την ε, ορατότητά της στην προβολή με τους πολίτες. Διότι η επικοινωνία με την κοινή γνώμη είναι κάτι το απαραίτητο προκειμένου να πετύχουμε στόχους. Θα πρέπει να γίνει μια πρόθεση εντός περιορισμένου αριθμού στόχων και σκοπών που θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί από την κοινή γνώμη και θα πρέπει αυτή η ενημέρωση, η επικοινωνία να γίνεται σε τακτά διαστήματα. Επίσης θα θέλαμε να δημοσιοποιηθούν οι προσανατολισμοί που θα αναλάβουν τα κράτη. Ε, καταλήγοντας να πω ότι οι Υπουργοί Οικονομιών ε, γνωρίζουμε αυτήν την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την Εστρατηγική, αλλά έχουμε καταδείξει την απόλυτη διαθεσιμότητά μας για να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε τον προσδιορισμό αυτού του νέας μορφής διακυβέρνησης και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους δύο βασικούς στόχους αηφόρος ανάπτυξη και απασχόληση ε, ποιοτική και κατάλληλη. Έτσι η Ευρώπη θα γίνει το κέντρο της οικονομίας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και αυτό θα αποτελέσει μια νέα φάση στο ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουλης. Ευχαριστώ όλους σας. Ε, thank you very much. Ε, ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρα. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια που καταβάλατε για να έλθετε στη συνεδρίαση σήμερα. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να μείνετε περισσότερο μαζί μας, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ασχοληθείτε και με τα εθνικά θέματα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρένα και μετά στον κύριο Γιούργεν Στάρκ. Ελπίζω ότι ο κύριος Επίτροπος και ο κύριος Στάρκ θα μπορέσουν να παραμείνουν και για την συζήτηση. Κύριε Ρένα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Σάρον, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκλησή σας να συμμετέχω στην συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αισθάνομαι όντως ε, ότι είναι μεγάλη τιμή να μπορέσω να συζητήσω την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε αυτό το φόρουμ ευρωπαϊκών πολιτικών. Η παρουσία γνώσεων και τεχνογνωσίας ε, και εμπειρογνωμοσύνης ε, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα, τη μοναδική δυνατότητα να κάνουμε μια καλή συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όπως σας είπε η κυρία Σαλγάδο, μόλις επιστρέψαμε από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup. Είχαμε μαραθώνια συνεδρίαση πάνω από 24 ώρες και χαίρομαι που μπορώ να συζητήσω μαζί σας αυτά τα θέματα τώρα που είναι ακόμη πολύ καινούρια και φρέσκα. Όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας της Ευρώπης, είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση έχει αλλάξει πολλά και μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την οικονομική ανάπτυξη που είχε με τις τελευταίες δεκαετίες τη θεωρούμε δεδομένη. Και αυτό ισχύει και όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Μέσα σε δύο χρόνια η κρίση κατάφερε να εξαλείψει 20 χρόνια βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Τίποτα δεν είναι όπως πριν και είναι ανάγκη πλέον να κάνουμε αλλαγές γιατί η κρίση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές και φορολογικές μας πολιτικές. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να παραμείνουμε στα ίδια, πρέπει να κάνουμε βηματικές αλλαγές προκειμένου να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Άρα πρέπει να κινητοποιήσουμε κάποιες ε, ατμομηχανές της ανάπτυξης για την Ευρώπη του 2020 να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία, τις θέσεις απασχόλησης και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα. Άρα αυτό που θέλουμε είναι βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πέρα από την διόρθωση των διαρθρωτικών αδυναμιών των αγορών μας και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα επενδύοντας τη γνώση, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Ας σας δώσω εδώ κάποια παραδείγματα. Στην εκπαίδευση ένας βασικός στόχος για την Ευρώπη του 2020 είναι να αυξήσουμε την συμμετοχή στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή τα σχολικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται υπό σημαντική πίεση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές να αντιμετωπίζουν πολύ πιο γρήγορες αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας από ό,τι στο παρελθόν. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να προετοιμάζουν τους μαθητές να αναλάβουν θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Άρα η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να δώσει σημαντικά ωφέλη όσον αφορά την δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας. Δεύτερο παράδειγμα, πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, ειδικά στους νέους καινοτόμους τομείς οι ψηφιακές υπηρεσίες νέας γενιάς και οι τεχνολογίες ενέργειας είναι τέτοια παραδείγματα νέων ευκαιριών. Η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, δίνοντάς τους περισσότερες επιλογές, αλλά και για τις επιχειρήσεις αυξάνοντας το μέγεθος της αγοράς και μειώνοντας το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε πολλούς τομείς που έχουν αντίκτυπο στις online υπηρεσίες και το online εμπόριο. Για την Ευρώπη του 2020 έχουμε έναν περιορισμένο, επαναλαμβάνω, περιορισμένο αριθμό στόχων που θα έχουν σαφή αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση της Ευρώπης. Καταρχάς, εκπαίδευση και έρευνα. Δεύτερον, ενέργεια, κλίμα. Αυτούς τους στόχους θα τους συζητήσουμε και θα τους προσαρμόσουμε στις ε, ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους μέλους. Και αυτοί οι στόχοι θα μας δείξουν τι όντως έχουμε καταφέρει στο θέμα της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το σημαντικό επίσης είναι όλοι αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την Ευρώπη του 2020 τόνισα ότι είναι σημαντικό να έχουμε στρατηγική δύο πυλώνων. Ρεαλιστική στρατηγική με οικονομική επιτυχία η οποία όμως θα βασίζεται και στην, στα καλά δημοσιονομικά και στην κινητοποίηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι η βάση της πρότασης της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην Ευρωζώνη δείχνουν ότι είναι επίγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε την, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Χτες είχαμε τη συνεδρίαση του Eurogroup, σήμερα την συνεδρίαση του ECOFIN και στις δύο περιπτώσεις τα Συμβούλια ενέκριναν την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Είχαμε και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και έναν εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει προκειμένου να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο για μείωση κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες του ελλείμματος το 2010. Είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν οι φορολογικές ανισορροπίες και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα προκειμένου να επανέλθει σε τομέα, σε τροχιά ανάπτυξης η Ελλάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα αλλά και εμείς δεν έχουμε διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την οικονομική σταθερότητα σε όλη την Ευρωζώνη, χτες το Eurogroup επανέλαβε τη δέσμευσή του για συντονισμένη δράση αν χρειαστεί διευκρινίσαμε κάποια τεχνικά θέματα όσον αφορά αυτή την συντονισμένη δράση που θα ξεκινήσει άμεσα αν χρειαστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για συντονισμένη και υπό όρους δράση και βοήθεια πέρα από την άμεση διαχείριση της κρίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Η ελληνική κρίση και η συνέχεια της μας έδειξε ότι χρειαζόμαστε αυξημένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Αυτή την ανάγκη την είχαμε ήδη αναγνωρίσει και προβλέψαμε την κατάλληλη νομική βάση στην συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προετοιμάζουμε προτάσεις για την εφαρμογή του άρθρου 136 της συνθήκης. Και ο στόχος μου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ενδεχομένως μία πρόταση για αυξημένη για αυξημένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής εντός των επόμενων δύο εβδομάδων πριν τα μέσα του Απριλίου. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε την ύπαρξη μη διαχειριζόμενων δημόσιων ελλημάτων. Πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωζώνης και να μπορούμε να κάνουμε πιο ευρείες και πιο αυστηρές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά τυχόν διορθωτικά μέτρα. Επίσης, η οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή απέδειξε ότι η ο συντονισμός της πολιτικής δεν μπορεί να αφορά μόνο τα φορολογικά μέτρα, όσο και αν αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν και άλλες μακροοικονομικές ανισορροπίες που μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες τόσο για μεμονωμένα κράτη-μέλη όσο και για την Ευρωζώνη. Για παράδειγμα, η μειωμένη ανταγωνιστικότητα και τα ελλείμματα στους ισολογισμούς είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Ενώ ακόμη και κράτη-μέλη που έχουν ε, μεγάλο πλεόνασμα στον εμπορικό ισολογισμό τους μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Κάτι που μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη σε όλη την Ευρωζώνη ενδεχομένως. Κάτι που μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε αλλαγή φορολογική σε όλη την Ευρωζώνη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων για την αύξηση της απασχόλησης και για την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης καθώς και για την ανάπτυξη. Μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης του 2020, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου στην Ευρώπη τα κοινοβούλια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ως νομοθέτες και πολλές από τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση για την Ευρώπη του 2020 θα εξαρτηθούν και από τη δική σας συνεισφορά και συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ανάπτυξη παράλληλα με την καλύτερη δημοσιονομική πολιτική, θέτοντας σημαντικές προτεραιότητες, κάτι που θα απαιτήσει πραγματικές πολιτικές επιλογές. Κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με δική σας στήριξη. Ελπίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην στήριξή σας για την Ευρώπη του 2020. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Περνάμε στην τελική παρουσίαση τώρα αυτή τη στιγμή με τον κύριο Γιούργεν Στάκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλο προνόμιο να είμαι εδώ ανάμεσά σα σήμερα και να συζητήσω μαζί σας αυτό το πολύ θα έλεγα έγκαιρο θέμα τη πολιτική και στρατηγική μέχρι το 2020. Το θέμα το οποίο θα συζητήσω και θα θίξω τα επόμενα λεπτά είναι το πώς έχουν τα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης και τα θέματα των στρατηγικών διεξόδου από την κρίση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι από την Άνοιξη 2009 είχαμε κάποια μηνύματα σταθεροποίησης μηνύματα βελτιώσεων και στις ε, χρηματοοικονομικές αγορές και στην οικονομία γενικά. Από την άνοιξη του 2009 λοιπόν οι αγορές, οι συνθήκες στις χρηματοοικονομικές αγορές έχουν βελτιωθεί και η οικονομική ζωή έχει ξαναξεκινήσει στις περισσότερες ε, χώρες. Και έχουμε λοιπόν παρότι με μετριοπαθή τρόπο στις πιο πολλές ε, ε, προηγμένες οικονομίες από δραστικά μέτρα υποστήριξης βέβαια απέρευσε αυτή η κατάσταση παγκόσμια και ταυτόχρονα είδαμε περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και αυτό είναι πάλι καλά μαντάτα. Όμως υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ακόμα και παραμένουν κίνδυνοι όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα. Στον τομέα της ε, ζώνης ευρώ, πρόσφατες πληροφορίες ε, καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη βρίσκεται ευθυγραμμισμένη με τον οδικό χάρτη. Όμως, οι γενικέ αναδιατάξει ε, που είναι αναγκαίες πιθανώς θα επιβαρύνουν την ανάκαμψη μέσα στη χρονική συνιστόσα, καθώς επίσης και οι επενδύσεις όπως οι επενδύσεις και οι αγορές εργασίας και οι προοπτικές αυτές ουσιαστικά θα είναι μέτριες δεδομένης και της ε, ε, πίεσης στην ζήτηση και κατανάλωση. Και έτσι θα είναι άνηση η ανάπτυξη και το 2010 άνηση σε σχέση με χώρες τομεακά άνηση και χρονικά στην κατανομή της άνηση. Με τις προοπτικές λοιπόν που έχει, έχουν κατατιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ευθυγραμμισμένες με προοπτικές άλλων, χρηματο... Ε, άλλων θεσμικών οργάνων όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μέση ανάπτυξη το 2010 θα είναι περίπου 1%. Όμως θα ε, ε, επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του 2011. Όσον αφορά τον πληθωρισμό και τις πληθωριστικές πιέσεις ήταν χαμηλές τους πρόσφατους μήνες. 0,9% τον Φεβρουάριο και η προοπτική για τον πληθωρισμό ευθυγραμμίζεται επίσης με τις προοπτικές για την σταθερότητα των τιμών αναμένουμε ότι θα παραμείνει ο πληθωρισμός ε, μεσοπρόθεσμα στο 1% και ότι μέσω της πολιτικής μας θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα λόγω του πλεονάσματος ε, του ε, δυναμικού και της μετριοπαθούς ανάκαμψης. Και αυτά πάλι ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ουσιαστικά ισορροπείται η κατάσταση όσον αφορά τις, ε, τη σταθερότητα των τιμών και ας το πω αυτό με κάθε σαφήνεια, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να υπάρχουν είτε πληθωριστικές είτε <clears throat> στασιμοπληθωριστικές ε, τάσεις. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την νομισματική μας, τις νομισματικές μας αναλύσεις στην αξιολόγηση χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων ε, μέσω πρόθεσμα όσον αφορά και την, τις προοπτικές για την ανάπτυξη. Συνολικά και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερά αγκυρωμένες μέσα στο πλαίσιο του στόχου μας να τηρηθούν τα επίπεδα πληθωρισμού <clears throat> κάτω από το περίπου 2% μεσοπρόθεσμα. Όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, πήραμε θαραλέα γενναία δράση ανταποκρινόμενη στην κρίση όσον αφορά τις πληθωριστικές τάσεις ε, που είχαν σημειωθεί λόγω της αυξημένης ύφεση, μειώθηκαν τα επιτόκια σε 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ρεκόρ χαμηλού επίπεδου, σε χαμηλά επίπεδα που δεν είχαμε στο την πρόσφατη ιστορία όσον αφορά την Ευρωζώνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι αυτό το χαμηλό επίπεδο των κυριότερων επιτοκίων είναι η εύθετη κατάσταση και πολιτική. Επιπλέον, πέρα από τη μείωση επιτοκίων, εμείς για να ενδυναμώσουμε τις ε, προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και για να διευκολυνθεί η παροχή αυτών των δανείων στις αγορές, εισαγάγαμε και έναν αριθμό ασυνήθιστων έκτακτων μέτρων. Πράγματι, αυτά τα μέτρα βελτίωσαν τις οικονομικές προϋποθέσεις, ιδιαίτερα τις αγορές, ε, συνεισφέροντας σε καλύτερη ροή πιστώσεων και στα νοικοκυριά και στις εταιρείε και επιχειρήσεις που κατά τα άλλα ε, δεν θα είχαν αυτές τις πιστώσεις. Είδαμε λοιπόν ότι σε σχέση με τα χαμηλότερα αυτά επιτόκια και τα έκτακτα μέτρα είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευθυγραμμιζόμαστε έτσι με ε, τα στοιχεία εκείνα που σε σχέση με την σύγκριση των ιστορικών αυτών στιγμών όταν χαμήλωσαν τα, ε, μειώθηκαν τα επιτόκια, η πολιτική αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρω με τι προσδοκίε. Θα ήθελα να πω όμω αυτά τα σημαντικά μέτρα, παρότι είναι πολύ σημαντικά για να διασφαλίσουμε την βελτίωση των συνθήκων και να διευκολύνουμε την παροχή χαμηλότοκων δανείων, δεν ε, θα παραμείνουν ενισχύει περισσότερο από ό,τι αναγκαίο. Πρέπει να εξετάσουμε το phasing out, την λήξη, την εκπνοή αυτών των μέτρων. Και ήδη τον Δεκέμβριο 2009 τον αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη σταδιακή εξάλληψη αυτών των έκτακτων μέτρων. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Ο λόγος είναι ότι όσο το μακρότερο συνεχίσουν να ισχύουν αυτά τα μέτρα, αυτό θα ε, οδηγούσε σε κίνδυνο σημαντικών στρεβλώσεων στις ε, νομισματικές αγορές, στις οικονομικές αγορές και θα έδινε και τα λανθασμένα μηνύματα ως κίνητρα. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά τις βελτιώσεις ε, από τις, ε, σε σχέση με τις, τους δείκτες από την εαρινή αυτή επισκόπηση θα ξεκινήσει αυτό το phasing out των έκτακτων μέτρων που αποφασίστηκε το Δεκέμβριο. Και έτσι μακροπρόθεσμα αυτό που είχαν αποφασιστεί στο παρελθόν πιο μακροπρόθεσμα. Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην κανονική, ε, στον κανονικό κύκλο των τρίμηνων ε, επιθεωρήσεων. Θα συνεχίσουμε την διευρυμένη αυτή ε, προσπάθεια παροχής πιστώσεων και δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους ε, βραχυπρόθεσμα στις ε, οικονομικές ε, συναλλαγές. Και αποφασίσαμε επίσης δύο εβδομάδες πριν να το κάνουμε αυτό όσο θα είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου. Για τους επόμενους λοιπόν έξι μήνες αποφασίσαμε να παραμείνουμε στο πλαίσιο των τακτικών αυτών δραστηριοτήτων μας χρηματοδόνως υποστηρίζοντας τις κανονικές αυτές δραστηριότητες. Όπως είχαμε αποφασίσει και τον προηγούμενο Οκτώβριο, εν συνόψη λοιπόν η φερεγγιότητα, η ρευστότητα όπω απαιτείται θα διασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το οικονομικό σύστημα με σταθερά επιτόκια. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει την σταδιακή phasing out, εξάλληψη οποιονδήποτε έκτακτων μέτρων για την ρευστότητα, τα οποία πλέον δεν θα χρειάζονται, δεν θα είναι αναγκαία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η μεσοπρόθεσμο, ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός είναι σημαντική υπόθεση για να υλοποιήσουμε την εντολή μας ε, της νομισματικής σταθερότητας όσον αφορά τη ζώνη ευρώ ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και θα ήθελα να πω ότι το phasing out αυτό ε, γίνεται για να αποφευθούν κίνδυνοι σε σχέση με την νομισματική ε, σταθερότητα που θα μπορούσαν να αναδυθούν υστερότερα σε μια μεταγενέστερη φάση. Και αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο. Ταυτόχρονα λοιπόν όμω θα αποφύγουμε υπερβολικά πρώιμη διέξοδο από τα έκτακτα αυτά μέτρα. Μια και κάτι τέτοιο θα διακύβευε την εξομάλυνση των αγορών και την ανάκαμψη. Φυσικά από την άλλη πλευρά δεν γνωρίζουμε ακόμα σήμερα ποια θα είναι η ομαλότητα της κατάστασης μετά από αυτή την κρίση που περνάμε και περάσαμε. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ακόμα το σενάριο και το πλαίσιο εργασιών μετά την κρίση. Όμως, κάνοντας λόγο για το τελικό σημείο αυτής της φάσης ε, εξάλληψης των έκτακτων μέτρων, το λειτουργικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε πριν από αυτήν την ε, χρηματοοικονομική κρίση τον Αύγουστο 2007 δίνει καλούς όρους και προϋποθέσεις ως γνώμονες. Και αν επιστρέφαμε σε αυτό το πλαίσιο πριν από την κρίση μόνο πολύ λίγες ε, παράμετροι της πολιτικής ε, θα ε, παραμείνουν όσον αφορά την διαδικασία υποβολής προσφορών όσον αφορά για παράδειγμα τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στις οποίες αναφέρθηκα μόλις πριν. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πολύ σύντομα στο γεγονός ότι πρόσφατα ακούστηκαν κάποιες φωνές και επιχειρήματα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα έπρεπε να αναλάβουν δράση ως διαχειριστές κινδύνων για να αποφευθούν συμβάντα και γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποπληθωρισμό σε στασιμοπληθωρισμό. Χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι θα έπρεπε να χαλαρώσουν οι στόχοι των κεντρικών τραπεζών και ότι θα έπρεπε να έχουμε στόχο υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Ω προ αυτά τέθηκε το θέμα αν δεν θα ήταν εύθετο να έχουμε διαρκώ υψηλότερους στόχους όσον αφορά τον πληθωρισμό τέθηκε η πρόταση και συζητήθηκε του 4%. Αυτό θα άφηνε μεγαλύτερο περιθώριο ώστε η νομισματική πολιτική να μπορέσει να αντιδράσει σε μεγαλύτερα και θα έλεγα ε, αντίξωα τέτοια φαινόμενα ή πλήγματα. Εγώ θα έλεγα ότι κάποια τέτοια αλλαγή θα ήταν σημαντικό σφάλμα. Σίγουρα μπορεί να είναι θελκτικό για κυβερνήσεις να προτείνουν υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού ώστε να δραματοποιηθεί η ε, κατάσταση όσον αφορά το ε, δημόσιο χρέος. Όμως, μια τέτοια κατάσταση αύξησης του ποσοστού πληθωρισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζει το κυριότερο πρόβλημα, το ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή <clears throat> θα είχαμε ανέφικτες ε, ε, πολιτικές ε, που θα αποτελούσαν ένα κίνδυνο μακροπρόθεσμα μέσα στο μακροοικονομικό πλαίσιο για την μακροοικονομική σταθερότητα. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι θα μπορούσε να απολέσει το κοινό οι πολίτες την γενική εμπιστοσύνη που έχουν όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του χρήματος, πράγμα το οποίο θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης όσον αφορά τις διαφορετικές προοπτικές για τον πληθωρισμό και αβεβαιότητα για τους επενδυτές. Αυτό ε, συνεπάγεται κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα θα συνέβαινε μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλότερων ποσοστών ε, πληθωρισμού. Θα έπρεπε εδώ να δούμε το ότι εμπειρικά στοιχεία επαληθεύουν ότι υπάρχει αρνητικό συσχετισμό μεταξύ αυτών των στοιχείων. Η νομισματική λοιπόν σταθερότητα υπονομεύεται εδώ διτά όσον αφορά την ε, ε, αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων έγκαιρα και δεύτερον όσον αφορά τις προσδοκίες ε, που θα πέραν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προστάτευε εν πάση περιπτώσει τις αγορές και τους ατομικά εμπλεκόμενους επενδυτές και έτσι θα ενθαρρύναμε υπερβολική ανάληψη κινδύνων από πλευρά τους. Αυτό με οδηγεί στα θέματα της φορολογικής πολιτικής. Πάλι σαν αντίδραση στην ε, οικονομική ε, κρίση και στην πρόληψη οικονομικής κρίσης στο ε, μέλλον. Θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα της sovereign debt crisis. Πολλές χώρες της ζώνης ευρώ αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα και δημόσιο χρέος. Ενώ, <clears throat> όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε η την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκτακτα μέτρα φορολογικίας ε, ε, αναλήφθηκαν και έπρεπε να αναλυθούν για να αποφύγουμε μια κρίση παρόμοια με του 1930 κρίσιμο στοιχείο σε σχέση και τώρα με την οικονομική ανάπτυξη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει σίγουρα αρνητικές παράπλευρες επιπτώσεις ε, για την ε, οικονομική ανάκαμψη. Θα ήθελα να πω ότι ε, μη εφικτές φορολογικές πολιτικές περιπλέκουν τα θέματα νομισματικής πολιτικής και το θέμα του έργου των, ευρωπαϊκών, των κεντρικών τραπεζών. Δημιουργούνται αβεβαιότητες και δημιουργείται ένα ρευστό πλαίσιο μεσοπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν η προοπτικές αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ε, επιβάρυνση των ε, σαντικές επιπτώσεις για τις επενδύσεις. Έχοντας εδώ τους ε, σταθεροποιητές που θα μπορούσαν να αναλειτουργήσουν ή κατά την διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων ανάληψη μέτρων, πραγματικά πολλαπλασιαστές ε, fiscal multipliers μπορούν να έχουν αντική επίπτωση και μπορεί να χρειάζονται προληπτικά ισχυρότερα μέτρα και έτσι να σημειωθεί συρρήκνωση οικονομική. Και πάλι αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του να μειωθούν τα επίπεδα χρέους και να έχουμε αποτελεσματικά μέσα και εργαλεία για να υπάρξει ισοστάθμιση, αντιστάθμιση στο μέλλον. Σαν αποτέλεσμα των ε, χαλαρώσεων των μέτρων μέσα στο πλαίσιο αυτό, πολλές χώρες της ζώνης ευρώ θα χρειαστεί να εμπλακούν σε μια φιλόδοξη πολιτική παγίωσης και σταθεροποίησης στο φορολογικό επίπεδο και να δούμε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στο 60% του ΑΕΠ τους όσον αφορά την επιβάρηση του, ε, ε, του, ε, του χρέους τους. Επιστρέφοντας τώρα σε σχέση με το θέμα της, από την κρίση, αυτό περίπου υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Κανένα σενάριο πολιτικής ή καμία προσαρμογή ή καμία παγίωση με άλλα λόγια θα οδηγήσει το χρέος σε πάνω από τα 100% του ΑΕΠ στη ζώνη ευρώ το 2015, σε 120% το 2020 και σε 150% το 2026 αν δεν ληφθούν μέτρα. Γι' αυτό είναι σωστό να διασφαλιστεί το θέμα της ρευστότητας. Για να διασφαλιστεί η ρευστότητα και η ε, αηφορία όσον αφορά τις φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να οδηγήσουν όλα αυτά στις κυβερνήσεις να θέσουν ως ανώτατη προτεραιότητα την φορολογική σταθεροποίηση και να φτάσει το επίπεδο της ε, <clears throat> το επίπεδο τους κάτω από το 3% όσον αφορά και τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ. Γι' αυτό ταυτόχρονα θα πρέπει αυτή η παγίωση και σταθεροποίηση να δούμε ότι θα πρέπει να διαρκέσει αρκετά χρόνια σε κάποιες χώρες, ώστε είτε το δημόσιο χρέος είτε το έλλειμμα να μπορέσουν να βρεθούν μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Το Σύμφωνο Ανάπτυξη και Σταθερότητα δίνει το εύθετο πλαίσιο για το συντονισμό των αναγκαίων πολιτικών σταθεροποίηση. Τώρα έχει φλέγουσα σημασία κυβερνήσει να έρθουν στο ύψο των περιστάσεων με τι υποσχέσει που είχαν δώσει, που πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειε αυτέ όπου είναι δυνατόν. Η κατάσταση αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει αυστηρή εφαρμογή αξιόπιστων κανόνων στο επίπεδο τη φορολογική πολιτική. Και τα πρόσφατα συμβάντα δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, να ενισχυθεί η εποπτεία, η επιτήρηση στην Ευρωζώνη και να εφαρμοστούν, να συμμορφώνονται όλοι με τους κανονισμούς. Αυτό με οδηγεί στην τελευταία μου παρατήρηση για την ανάγκη διαρθωτικών αλλαγών και προσαρμογών. Πολλά έχουν αναφερθεί από πλευράς Προέδρου και Επιτροπής. Όμως θα ήθελα αυτά να τα θέσω στο σωστό πλαίσιο. Η, η υγιής οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να ανακουφίσει την πίεση, μειώνοντας ε, ε, το την πίεση σε σχέση με την οικονομία και βελτιώνοντας τους αιτήσους προϋπολογισμούς στα δημοσιονομικά. Αυτό υπογραμμίζει πάλι τη σημασία του να υπάρξει άξιση του δυναμικού των οικονομιών μας. Όμως το σημείο φετηρίας η εκκίνησή μας δεν είναι η καλύτερη. Οι περισσότερες εκτιμήσεις από διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δείχνουν ότι έχει μειωθεί ταυτόχρονα και το επίπεδο και το ποσοστό ανάπτυξης ε, στην ε, ε, ανακαμψή μας. Είναι λοιπόν κέρια σημασία να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις που θα αναζωογονήσουν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάκαμψη και την απασχόληση. Πολιτική που θα αυξάνει την, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Επιγόντως χρειαζόμαστε αυτές τις πολιτικές για να επιταχύνουμε τις διεργασίες, να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, νέες ευκαιρίες του επιχειρήν και να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός σε εκείνες τις περιφέρειες και χώρες που δεν είναι ε, ανταγωνιστικές ακόμη και που περιφέρειες έχουν ολόκληρες χάσει την ανταγωνιστικότητά τους ε, ε, το τελευταίο διάστημα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η αναδιάταξη, η αναδιάρθρωση και του τραπεζικού τομέα, βελτίωση των ισολογισμών, βελτιωμένη διαφάνεια έχουν πολύ μεγάλη σημασία επίση. Ολοκληρώνω, επιτρέψτε μου, πρώτον, η παγκόσμια οικονομία δείχνει κάποια μηνύματα διαρκέστερη ανάκαμψη. Στην Ευρωζώνη επίση βρισκόμαστε καθοδόν προ την ανάκαμψη, παρότι με ένα πιο μέτριο ρυθμό και οι αβεβαιότητε παραμένουν υψηλέ. Δεύτερον, όσον αφορά τι νομισματικέ μα πολιτικέ, εξακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε το παρόν επίπεδο των ε, κύριων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως ε, σωστά μέτρα δεδομένου του ε, των χαμηλών, δεδομένων των χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων και της νομισματικής σταθερότητας. Οι βελτιωμένες αυτές καταστάσεις όσον αφορά ήδη την άνοιξη του 2009 μέχρι σήμερα δείχνουν ότι είναι ανάγκη να εξαλειφθούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από πλευράς μας υπάρχει ανάγκη να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναγκαίο. Τέταρτο, αυτό δεν σημαίνει όμω ότι η κρίση ολοκληρώθηκε και έχει περάσει. <clears throat> Μπορεί να υπάρξουν ε, κάποιε αντικσοότητε, μπορεί να υπάρξουν μελλοντικέ προκλήσει ε, και πρέπει εδώ πραγματικά να είμαστε προετοιμασμένοι και η περίπτωση τη Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι πρέπει να ε, τελούμε ενεγρηγόρση. Δεύτερον, οι, οι κεντρικές τράπεζες θα έπρεπε να δώσουν τα αναγκαία μέτρα για την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη και να πάψει να υπάρχει οποιαδήποτε βεβαιότητα προς την λαθασμένη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδηστε η συνεδρία σε αυτή να γίνεται παράλληλα με την συνάντηση ε, του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά αυτό έχει ως επιπτώσει να μην μπορούν να παραστούν κάποιοι του συγκεκριμένου μα. μας. Θα συνεχίσουμε τώρα με την συζήτηση, διότι θεωρώ πως θα πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων και θα καλέσω τον κύριο Στάρκ να απαντήσει ενδεχομένω σε ερωτήσεις που θα του τεθούν. Έχουμε και τον κύριο Σανοφέρη εδώ που ίσως ε, και αυτός θα μπορούσε να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που ενδεχόμενα να του φανούν ενδιαφέροντα. Θα σας πω το κατάλογο των αγοριτών που έχω μαζέψει μέχρι τώρα. Got... Από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω τα ονόματα. Sorry, the, from Italy, uh, Mr. Angelo Ferrugia from Malta and uh, Mrs. Person Peterson from Latvia and from the European Parliament I've got Jose και από το Ευρωκοινοβούλιο, τον Μαγκάγιο. Sven Giegold, Edward Sikluna and Adi Podimata. Um, if there's anybody else who... Αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να προσθέσουμε το όνομά του, παρακαλώ, κάντε ένα νεύμα. Η γραμματεία φροντίζει να πάρει τα ονόματά σας. Γερουσιαστής Ντεμπρόφσκι από την Πολωνία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης η Πολωνία τα πήγε σχετικά, θα λέγαμε αρκετά καλά. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που σημείωσε οικονομική ανάπτυξη το 2009. Παρότι αυτή η ανάπτυξη ως ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι πριν από την κρίση. Επίσης είμαστε επιτυχείς χάρη στα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει για να αντισταθμιστούν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Παρόμοια μέτρα με αυτά τα οποία υιοθέτησαν άλλες χώρες βέβαια. Αύξηση των εγγυήσεων κεφαλαίων των καταθέσεων κεφαλαιακών εγγυήσεων, η αποταμίευση όσον αφορά εξοικονόμηση δαπανών σε σχέση με τον δημόσιο τομέα, κινητοποίηση των, της υποστήριξης όσον αφορά την εξόφληση υποθηκών ε, η βοήθεια όσον αφορά δάνεια και πιστώσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθιστώντας ε, πιο εύκολο το πλαίσιο δανεισμού για αυτές ε, ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την κρίση και συναφή θέματα μέτρα επίσης για την προαγωγή θέσεων απασχόλησης όσον αφορά την αγορά εργασίας και απασχόλησης μέτρα προς όφελος και των εργαζομένων και των εργοδοτών βέβαια. Τα κάναμε όλα αυτά με νομοθετικό έργο το οποίο αναλάβαμε ως πρωτοβουλία. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών σταθεροποιήθηκε η πολωνική οικονομία. Επετέχθη λοιπόν σταθεροποίηση. Και η Ευρώπη οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι Κίνα, η Ιαπωνία, όλες αυτές οι χώρες πρέπει να αναλάβουν μέτρα και εκείνες η Ευρώπη όμως υποφέρει από υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος το οποίο παρακολεί την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης η Ευρώπη έχει επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την έκκληση των αερίων διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αυτό είναι εξόφθαλμο και ιδιαίτερα διάκριτο για την Πολωνία που εκμεταλλεύεται τον λιθάνθρακα και όλα αυτά από την άλλη πλευρά οδηγούν σε επιβάρυνση του κόστους ενέργειας παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη συνολικά. Αυτού του είδους τα μέτρα δεν υπάρχουν όμως σε άλλες χώρες, δεν υιοθετούνται από αυτές. Και έτσι σαν αποτέλεσμα τούτου αυτή η μονοβαρής διαμόρφωση των συνθήκων ανταγωνισμού δημιουργεί αρνητικό περιβάλλον για την Ευρώπη γενικά. Μέχρι σήμερα σε σχέση με την ε, επιβάρηση του κλίματος από το διοξίδιο του άνθρακα πιστεύω ότι όταν υπάρχουν ε, ενδείξεις για μια αρνητική επιβάρηση του κλίματος οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν ισομερώς παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα, οικουμενικά. Στην Πολωνία, στην περιοχή Μπελγκάντοφ όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό τον σταθμό έχουμε σύλληψη άνθρακα και αποθήκευση άνθρακα αποθήκευση άνθρακα υπόγεια αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα παραγωγής ενέργειας αυτού του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% αυτό σημαίνει αυξημένη καύση άνθρακα αυξημένη έκκληση αερίου, αερίων διοξιδίου του άνθρακα και σύλληψη και αποθήκευση αυτού του διοξιδίου του άνθρακα υπόγεια. Δεν μπορώ να δω πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί κερδοφόρο μακροπρόθεσμα. Ο εντόπιος επιτόπιος πληθυσμός επίσης ανησυχεί για τις περιβαλλοντικά αρνητικές επιπτώσεις που θα συνεπαγόταν αυτή η σύλληψη και αποθήκευση υπόγεια του άνθρακα, του διοξιδίου του άνθρακα θα έπρεπε σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Βοημίας και της δασόδης μας περιοχές να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία αν συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί. Ένα άλλο θέμα, ε, ε, το επισητιστικό θέμα η παραγωγή τροφίμων. Έχουμε μεγάλε εκτάσει στην Πολωνία που είναι χέρσες και δεν καλλιεργούνται. Όμω αυτό πρέπει να το δούμε σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων. Δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά στην καλλιέργεια, διότι δεν υπάρχει καμία, καμία επιστημονική ένδειξη που να αποδεικνύει ότι αυτά είναι ασφαλή. Πολλέ φορέ γίνεται λόγο, βέβαια για τα περιβαλλοντικά θέματα και την υγεία, αλλά πολύ λίγα μα λένε όσον αφορά τι πιθανέ αρνητικέ επιπτώσει ε, που μπορούν να έχουν όλα αυτά στη δημόσια υγεία. Κάποια είδη δηλαδή τροφίμων. Θα πρέπει να προάγουμε την υγιή διατροφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια δεν νομίζω ότι ακούσαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά ακούσαμε μια σύνοψη της κατάστασης στην Πολωνία που ήταν επίσης χρήσιμη. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πιο συντηρητικοί στο χρόνο που χρησιμοποιούμε. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Ιταλικής Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θέλω λοιπόν να υποστηρίξω την Ιταλική εργασία και άρα θα περάσω στην Ιταλική. Ευχαριστώ. Πιστεύω πως ε, για μια στρατηγική ανάκαμψης, ε, ανάπτυξης και απασχόληση μέχρι το 2020 χρειάζεται να κατανοήσουμε απολύτως ε, ποιε ήταν οι αιτίε αυτής της κρίσης που διανύουμε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ανάκαμψης ε, της παραγωγικής δραστηριότητα ε, την οποία γνωρίζουμε σήμερα. Διότι αν ε, δεν τα κατανοήσουμε όλα αυτά, πολύ νωρίτερα από το 2020 θα ξανααντιμετωπίσουμε μια μεγάλη σοβαρή παγκόσμια κρίση. Οι τρεις αιτίες της κρίσης που ζήσαμε αλλά και που συνεχίζουμε να ζούμε είναι πρώτον η πραγματική ανισορροπία που υπήρξε στην παγκόσμια οικονομία. Η υπερβολική κατανάλωση από πλευράς Αμερικανών, η υπερβολική, ε, υπερβολική ε, επενδύσεις από πλευράς ε, Κίνας και η αποταμίευση και η συμπεριφορά της Ευρώπης, κάτι το οποίο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύσσεται με ποσοστά λιγότερο το 1% τα τελευταία χρόνια πριν από την κρίση, δηλαδή το 1 τρίτον των ΗΠΑ και 1 τέταρτον των 5 της Κίνας. Ο δεύτερος λόγος ήταν η έλλειψη κανόνων στις χρηματαγορές και ως εκ τούτου η δημιουργία των περίφημων ε, φουσκών και η τρίτη αιτία είναι η ακαταλληλότητα μιας παλιάς διακυβέρνησης του παλιού G8 ενώπιον του νέου κόσμου. Άρα λοιπόν μια, η απέτηση για μια νέα μορφή διακυβέρνησης. Αν λοιπόν δούμε τα σημάδια της ε, μεγέθυνσης της ε, διεθνούς οικονομίας, αυτά τα σημάδια βασίζονται στις τρεις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση. Δηλαδή, η ανάκαμψη στηρίζεται στην υπερβολική κατανάλωση των ΗΠΑ, στην αποταμίωση των Κινέζων, δεν υπάρχουν νέοι κανόνε στο διεθνέ ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν έχει προκύψει ακόμα μια νέα διακυβέρνηση. Ο κόσμο λοιπόν βρίσκεται σε, μια είδος, ένα impossibility theorem που πριν από 50 χρόνια ο οικονομολόγος Kenneth Harwood ανέφερε για να θίξει άλλα ζητήματα, άλλα προβλήματα. Αλλά σήμερα η κατάσταση αυτή οφείλεται σε τρεις μεγάλες περιοχές, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, Ευρώπη και ε, η Ιαπωνία, πιστεύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν την κρίση χρησιμοποιώντας ε, το μοντέλο του export-led, δηλαδή να, κατευθύνει, να κατευθύνει τα πράγματα ή το εξαγωγικό εμπόριο αλλά κάθε πλευρά από τις τρεις πιστεύει ότι μπορεί να εξέλθει από αυτή την κρίση στηριζόμενη και βαζόμενη στις εξαγωγές, το ερώτημα είναι απλό. Ποιος αγοράζει αυτές τις εξαγωγές, αυτά τα προϊόντα και πώς μπορούμε να εξορροπήσουμε τις πραγματικές ανισότητες που υπάρχουν στην πραγματική οικονομία και εν τέλει στο θεώρημα της ε, αδυναμίας ε, αυτή τη ε, παγκόσμια οικονομία υπάρχει η ωραία κοιμωμένη του δάσου που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν έχουμε ανάγκη από μια νέα διακυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε μια διακυβέρνηση με ένα G20, G25, G30. Πρέπει να έχουμε ένα νέο G8, μια λέση των 8, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν η Ινδία, η Ιαπωνία, οι Πολιτείε, η Ρωσία, η Βραζιλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη είτε θα είναι παρούσα στην νέα διακυβέρνηση με τα Ηνωμένα κράτη της Ευρώπης ή δεν θα είναι παρούσα καθόλου διότι αυτά τα, αυτές οι οντότητες της νέας governance θα πρέπει να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομικού συστήματος ένα νέο Bretton Woods την ε, βασική αναθεώρηση του ε, διεθνούς ε, Οργανισμού Εμπορίου, του παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου. Δηλαδή δεν μπορεί να εισέρχεται ε, η Κίνα σε ένα τέτοιο οργανισμό ελεύθερα, αλλά να ε, κάνει ε, να ασκεί πιέσεις στο δολάριο απ' την άλλη. Αυτό το οποίο βλέπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έλλειψη ενός στρατηγικού πλαισίου για μακροοικονομικές πολιτικές σε σχέση με τις οποίες οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες άκουσα να αναφέρονται στις εισαγωγικές ομιλίες, όλα είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Ευελιξία στην αγορά εργασίας, αυστηρότητα από πλευράς ε, χρηματοπιστωτικής, κινδυνεύουν κατά την άποψή μου να μη σημαίνουν τίποτα, εν, ε, απουσιάσει ένα πλαίσιο αναφοράς για ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης, δηλαδή ένα εφόρο σύστημα σε ε, παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να περάσει στο Μάστριχ 2 αφενός, περισσότερη αυστηρότητα, λιτότητα, όχι ε, ελλείμματα και επενδύσεις σε θέματα υποδομών, καινοτομίας, νανοτεχνολογιών κλπ. Όλα αυτά αναφέρθηκαν και ένα νέο καθεστώς για την ευρωπαϊκή ε, κεντρική τράπεζα που δεν θα την περιορίζει μόνο στον έλεγχο του πληθωρισμού και των πιέσεων, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις παλάπλευρες επιπτώσεις που η υπερεκτίμηση του ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση των ποσοστών ανάπτυξης. Χρειάζονται δύο σκέλη για την μισονική πολιτική. Ανάπτυξη και και για την φορολογική πολιτική χρειάζεται μεγαλύτερη αυστηρότητα, μεγαλύτερη λιτότητα, ε, ε, ένα πλεόνασμα των ε, εθνικών προϋπολογισμών αλλά και ανάπτυξη παράλληλα. Το ερώτημα έχει ως εξής τι ομιλούμε σε αυτές τις συζητήσεις μας όταν βάζουμε τον τίτλο «Στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση μετά την κρίση και την έξοδο από την κρίση του 2020» εάν μεταξύ βλέπουμε ότι η οικονομία προχωράει προς μια νέα μεγάλη κρίση ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης για να αποφύγουμε και να προλάβουμε μια τέτοια υπόθεση και να συμβάλλουμε στο νέο ε, οικονομικό και νομισματικό παγκόσμιο γίγνεσθε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έβαλα μπροστά το ρολόι διότι πρέπει να λάβετε το λόγο λιγότερο από τρία λεπτά, διαφορετικά ε, οι συνάδελφοι θα αρχίσουν να σας ε, μαχαιρώνουν πισόπλατα στο δείπνο απόψε. Ε, κοιτάξτε, σας υπενθυμίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, συζητήσουμε τις σφαιρικότερες πτυχές της εξόδου από την κρίση αύριο. Τώρα περνάω στους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο. Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δράτοντας την ευκαιρία που βρίσκονται εδώ ο κύριος Στάρκ και ο κύριος Πιζανή θα θέσω ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Κύριε Στάρκ, τι γνώμη έχετε για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για το οποίο συζητάμε. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Η στρατηγική για το 2020 περιλαμβάνει και μία παράγραφο που λέγεται ότι λαμβάνουν υπόψη την ευθύνη του ε, χρηματοπιστωτικού κλάδου στη συμβουλή στην κρίση θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιους μηχανισμούς που θα ε, τους έκανε να πληρώσουν το κόστος αυτής της κρίσης. Αυτή η δήλωση δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται με τις προτάσεις της Κομισιόν ούτε του Συμβουλίου σε ζητήματα εποπτείας των τραπεζών. Το Κοινοβούλιο πρότεινε ένα μηχανισμό παρόμοιου τύπου για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα τη στρατηγικής 2020. Ε, με εκπλήσει που το Συμβούλιο όταν ε, το ακούσαμε χθε δήλωσε ότι είναι κατά της ιδέας αλλά και την ίδια στιγμή εγκρίνει κάτι παρόμοιο στο πλαίσιο στρατηγικής 2020. Και στο κύριο Πιζανή μια ερώτηση πολύ σύντομη. Ε, στο Στρασβούργο ο Πρωθυπουργό τη ε, Ισπανία μιλούσε για ένα σύστημα για την πολύ κυρίσεων. Στη το 2020 μιλάει μόνο για το άρθρο 121, μεγάλου προσανατολισμού και φυσικά συντονισμό στον χώρο του ευρώ, όπω ε, δήλωσε και η Προεδρία. Είναι κάτι που ήδη γνωρίζαμε όταν ο Πρόεδρο ε, έκανε αυτή την πρόταση. Πρόεδρο του Συμβουλίου. Μπορείτε να προβλέψετε ποια είναι η προσθέμενη αξία που η Ισπανική Προεδρία θέλει να προσθέσει στα άρθρα αυτά τα οποία ήδη γνωρίζαμε με την πρόταση αυτή, διότι σε όλα τα έγγραφα βρίσκεται, βρίσκεται στο δανεικό κείμενο, στο ιταλικό, στο κείμενο της Βουλής των Λόρδων, ε, το θέμα της συζήτησης, ε, αυτή τη διακυβέρνηση που προς το παρόν δεν ε, έχει καταστεί τίποτα το σαφές και το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Θα ακούσω μερικές ερωτήσεις ακόμα. Κύριος Άντζελο Φρουίζη από την Μάλτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις παρουσιάσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση για το 2020. Όμως, με τη Μάλτα που είναι η μικρότερη οικονομία μεταξύ των 27 και που αυτή τη στιγμή έχει πολύ χαμηλές επιδύσεις στην εκπαίδευση με και βρίσκεται στην 60η θέση όσον αφορά την εκπαίδευση γενικά και στη θέση γύρω στο 50 όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, βλέπουμε ότι το ΑΕΠ μας είναι το 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η φτώχεια αυξάνεται δραματικά στη Μάλτα με πάνω από 20% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας και να πω ότι στη φτώχεια συμβάλλουν και οι μεγάλες αυξήσεις στο κόστος του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος που ήταν οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη των 27 με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Αυτή τη στιγμή 21% των παιδιών που ζουν στη Μάλτα βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, κάτι που οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης έχουμε μεγάλη αύξηση της ανεργίας καθώς και του ελλείμματος. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και την απασχόληση για τις μικρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν τόσο αποδοτικά οι ίδιες στρατικές που χρησιμοποιούνται για τις μεγαλύτερες γλώσσες. Ευχαριστώ και να σας προειδοποιήσω ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τη διερμηνία αν μιλάτε πολύ γρήγορα. Τώρα θα ακούσουμε κάποιες ακόμη ερωτήσεις πριν περάσουμε σε απαντήσεις. Από την Λετωνία, κυρία Πίτερσον. Ευχαριστώ. Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε και αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έδειξαν στη Λετωνία σε μια εξαιρετικά κρίσιμη οικονομική συγκυρία. Σήμερα όμως τι βλέπουμε 20% μείωση στο ΑΕΠ, 20% ανεργία, 30% μείωση των ε, αμοιβών στο δημόσιο τομέα και επίσης 30% μείωση στο λιανικό εμπόριο. Αυτά είναι τα στοιχεία για τη Λετωνία. Βεβαίως είναι καλό που η κρίση τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λετωνία δεν μας ανάγκασε να αλλάξουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Όμως αυτή τη στιγμή στη Λετωνία πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε διαφορετικές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Συζητήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους ε, στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα της Επιτροπής και καταλήξαμε στη συμφωνία ότι οι προτεραιότητες μας είναι οι εξής. Μαϊκρονομική σταθερότητα, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση. Πέρα όμως από αυτό μας ενδιαφέρει και οικονομική πέρα από την κοινωνική συνοχή. Τι εννοούμε με αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει στήριξη στις ε, περιοχές της υπαίθρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει μια ισότιμη μεταχείριση όλων των φορέων που συμμετέχουν στον γεωργικό τομέα και εξισορρόπηση των άμεσων ενισχύσεων. Ειδικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη στις πιο φτωχές, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε το βασικό στόχο της στρατηγικής που είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης πολιτικής οικονομίας της, αγορα... της κοινωνικής αγοράς. Βλέπουμε φιλόδοξους στόχους στη στρατηγική. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να πιέσετε το χρόνο, αλλά μιλάτε πολύ γρήγορα. Αν μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο σιγά οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να είναι τέτοιου είδου, ώστε να είναι πραγματικά να επιτευχθεί η εφικτότητα, να είναι εφικτή. Και θα είναι πιο ρεαλιστικό αν θα καταφέρουν τα κράτη-μέλη να ποσοστοποιήσουν του στόχου του ευθυγραμμιζόμενα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Θα θέλαμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ΜΜΕ, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να δουλέψουμε με νομοθεσία υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τώρα πολύ σημαντικό αυτό μέσω τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν είναι σαφέ ποιε θα είναι οι προτεραιότητε αυτή τη στρατηγική για το 2020 και πώ θα συνδέονται με τα δημοσιονομικά, με τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαθωτικά ταμεία. Ποιο θα είναι το ποσοστό του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού του στόχου και ποιε θα είναι οι απαιτήσει και εν τέλει κάποιες συστάσει από πλευρά μου. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει άντληση κονδυλίων από διαφορετικές πηγές και όχι μόνο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν έξι λεπτά, λέγει η Πρόεδρος. Και πολλοί άλλοι θέλουν να παρέμουν μετά από εσά. Μπορείτε να ολοκληρώσετε. Για να ολοκληρώσω, λέει ο Μιλητρία, θα ήθελα απλά να πω ότι προτείνουμε να αξιολογηθεί αν η πρωτοβουλία αυτή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκαία για αυτή τη στρατηγική. Νομίζουμε ότι αν με επιτυχία καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους έξι, τις έξι πρωτογενείς πρωτοβουλίες τότε το ε, πρόβλημα παίρνει άλλες διαστάσεις. Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συντονισμό των προσπαθειών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι να υπάρξει μια παρουσίαση αποτελεσματική αυτών των θεμάτων από πλευρά ε, των κρατών και της Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κατανοώ ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Ζητώ από όλου σα να προσπαθήσετε να είσαστε συντομότεροι στις παρεμβάσει σας. Φιλίπ Λαμπέρτ στη συνέχεια. Παρακαλώ, Φιλίπ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πειθαρχημένο. Πρώτον, εκφράζω την θλίψη μου για το γεγονό ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποχώρησαν. Δεν είναι μήνυμα σεβασμού προ του εθνικού εκπροσώπου βουλευτέ, που μια φορά κάθε τόσο έρχονται σε εμά για να συμμετάσχουν εδώ σε αυτέ τι εργασίε. Έχω κάποια πράγματα να πω για το 2020, μια όμω και ο επίτροπο αποχώρησε, θα το αφήσω για ιστερότερα για άλλη φορά. Πρώτον, για την παραγωγικότητα. Αναφέρθηκε πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Για ποια παραγωγικότητα κάνουμε λόγο, για την εργασιακή παραγωγικότητα τη εργασία, αν είναι αυτό τότε αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να αυξηθεί η οικονομία θα πρέπει να αυξηθεί και το αποτέλεσμα παραγωγικότητα, παραγωγικότητας από πλευράς των εργαζομένων μας. Και αυτό είναι κάτι το ανέφικτο. Λοιπόν, κύριε Στακ, κύριε Πιζανή Φερή, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση από αυτόν. Διότι θεωρούμε ότι εδώ είναι μια, ας το πω έτσι, μη ίση εξίσωση εδώ. Δυσανα... Ε, μη εξισορροπημένη εξίσωση. Θα ήθελα να πω για την φορολογική πολιτική. Ακούμε υπερβολικά πολλά πράγματα για τη φορολογική σταθεροποίηση όσον αφορά τον τομέα των δαπανών, την χρηματοοικονομική πολιτική για τι δαπάνε. Δεν ακούμε πολλά για τα έσοδα. Τι κάνουμε δηλαδή με το σύστημα φορολόγηση και τα φορολογικά έσοδα, ώστε να καταφέρουν οι κυβερνήσει μα να παράσχουν τι υπηρεσίε που πρέπει να παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να μεταθέσουμε το κέντρο μέτρο των φορολογικών πολιτικών μα και των συστημάτων μα ε, φορολογικών εσόδων για να είναι πιο αποτελεσματικά. Και τι θα γίνει σε σχέση με τα έσοδα τα οποία χρειάζονται τα κράτη-μέλη για να παράσχουν αυτέ τι υπηρεσίε. Τρίτο, οι ανισότητε. Ακούμε πολλά σχετικά για τι ανισότητε στου τρέχοντε λογαριασμού κτλ. Υπάρχει μια ανισορροπία που θα ήθελα να τοποθετηθείτε επ' αυτή ε, όσον αφορά το πρόβλημα τη φτώχεια. Έχουμε 16% φτώχεια στην Ευρώπη που πρόκειται για μια προηγμένη οικονομία όπως την αποκαλούμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε ποιο βαθμό είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ανέφικτο ως ανισότητα αυτή την κατάσταση. Είναι ένα ευκταίο αποτέλεσμα της πολιτικής μας ή είναι ένα αίτιο, μια από τις ρίζες ε, των, ε, του, το, της κακοδαιμονίας μας αυτής της κρίσης. Αν είναι ένα αίτιο, μια ρίζα, ε, τότε δεν είναι για φιλαλληλία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι και για οικονομικούς λόγους και λόγους αποτελεσματικότητας που πρέπει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Πώ το βλέπετε, είμαι κάτω από τρία λεπτά στο χρόνο παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Περνώ τώρα και στρέφομαι σε εσά. Ή όχι, θα έχουμε τον γύρο απαντήσεων τώρα μετά από αυτέ τι παρεμβάσει, γιατί θα ξεχάσετε αλλιώ τι ερωτήσει που διατυπώθηκαν. Έχουμε που διατυπώθηκαν προς εμάς. Δεν ξέρω, θέλετε εσείς να τοποθετηθείτε τώρα και μετά στη συνέχεια θα περάσω ε, σε εσάς Σταρκ. Εσείς έχετε πρώτος τον λόγο, παρακαλώ. Όπως ε, προφανώς αναφέρθηκε, είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένο που είμαι εδώ ανάμεσά σας και έχει προσφερθεί αυτή η ευκαιρία σε, σε μένα να ε, συζητήσω αυτά τα θέματα μαζί σας. Πρώτα θα ήθελα να απαντήσω τη δική σας ερώτηση για τις κυρώσεις και για την δυνατότητα χρήσης κάποιας μορφής κυρώσεων για να επιβληθούν οι στόχοι και να συμμορφωθούν όλοι με τους στόχους της ημερησίας διάταξης ατζέντα για το 2020. Η προσωπική μου άποψη για τις κυρώσεις είναι, όπως είδαμε με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθούν και να εκτελεστούν οι κυρώσεις αυτές. Ουσιαστικά ο λόγος είναι ότι μόνο τότε κυρώσεις μπορούν να εξεταστούν όταν θα έχει αποδειχθεί. Θα είναι δεδομένο ότι η συμπεριφορά μιας τάσης, η τοποθέτησή, σας, τοποθέτησή της έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, όχι μόνο για αυτή την ίδια αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ κτλ. Αυτός είναι ο μόνος ε, σκόπιμος λόγος για την επιβολή κυρώσεων. Κατά τα άλλα, πολιτικά και διεθνώς δεν είναι κάτι το εφικτό να εξετάζει κανείς επιβολή κυρώσεων για άλλους λόγους. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, οποιοδήποτε κι αν είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι θέμα ουσίας αυτό, εντάξει. Τώρα για την ίδια την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά το νέο πλαίσιο πολιτικής, New Policy Framework, όπως συζητείτε για την πολιτική της ΕΕ μέχρι το 2020 και το θέμα των προσαρμογών μέσα στη ζώνη ευρώ, με την έμφαση στον συντονισμό φυσικά. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο ποιο είναι. Έχουμε μια νομική βάση η οποία δεν προβλέπει όμως κυρώσεις έχουμε μια νομική, ένα νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποβολή συστάσεων. Το γεγονό ότι κατά το παρελθόν δεν έγινε χρήση των συστάσεων αυτών ώστε να κατανοήσουν οι κυβερνήσει ότι οι εξελίξει στη χώρα του ε, ήταν αρνητικέ και δημιουργούσαν προβλήματα, ένα, ένα θέμα μη μη επίτευξη στόχων για την ίδια τη χώρα και για την ΕΕ. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και ως ε, μη, μη ε, δραστικό μέσο. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μη δραστικά μέσα εφόσον η έμφαση βρίσκεται στο να αποσαφηνίζεται πάντα και να διευκρινίζεται ποιες είναι οι απαιτήσει. και τι, πού δημιουργεί και πώς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά προβλήματα για τη σταθερότητα και την επίρρευση των στόχων. Αυτό που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και αναφέρομαι εδώ στην παρέμβαση του Ευρω... της, Ευρωβουλευτίνας, της ε, εκπροσώπου της ε, Λετωνίας ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσον αφορά την ενίσχυση, την ενδυνάμωση της κοινή δέσμευση για την επίτευξη κοινών στόχων μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής για το 2020. Αυτό ήδη είχε συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την συνθήκη της Αβώνας. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλύτερα η πολιτική του καρότου παρά της μαγκούρας, παρά του μαστίγιου. Να δίνουμε κίνητρα και όχι να έχουμε τόσο τιμωρίες και κυρώσεις. Τώρα, το άλλο για την πραγωγικότητα ως βάση για την αηφορία και την ανάπτυξη. Δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα ποσού, ε, όγκου της παραγωγικότητας ε, ως αριθμού. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας η παραγωγικότητα. Αν είσαστε αποτελεσματικοί, καλό αυτό. Δεν μπορείτε να εκφράζετε τη θλίψη σας για το γεγονός ότι είσαστε παραγωγικός. Το θέμα είναι τι παράγεται. Η αηφορία εκφράζεται πολύ περισσότερο υπό τους όρους του τι παράγεται και τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα με την οποία παράγεται αυτό το αγαθό σε σχέση με διάφορα άλλα αγαθά τα οποία επιθυμεί κανείς να έχει στην οικονομία του. Δεν είναι θέμα όγκου παραγωγής, έτσι. Δεν ε, πρέπει κανείς να κατηγορεί κάποιον ή να υπάρχει ενοχή για να είναι παραγωγικός. Εδώ παραγωγικότητα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και παραγωγικότητα όσον αφορά τους πόρους. Εδώ αυτό πρέπει να δούμε για διαφοροποίηση. Συμφωνώ μαζί σας λέει ο μιλητής ότι έχουμε εδώ μια προκατηλημένη ε, τοποθέτηση όσον αφορά την εργασιακή παραγωγικότητα. Δεν λαμβάνει υπόψη πόσο κεφάλαιο καταναλώνεται, πόσοι πόροι καταναλώνονται και αυτό πρέπει να βαίνει πάντα να ε, αναλογεί πάντα με το, την παραγωγικότητα του τελικού προϊόντος. Πρόκειται όμως για σωστή μέτρηση, για την θα έλεγε κανείς ανάλογη ορθή μέτρηση αντί να έχουμε μια ανώτατη οροφή απλώς συλλήβδην. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσείς κύριε Στάρκ. Thank you very much for the questions addressed. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Φοβάμαι ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν δεν είναι όλες ερωτήσεις που μπορώ να απαντήσω εξαιτίας της διαφορετικής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όσον αφορά το μακροοικονομικό πλαίσιο και τα διδάγματα που πρέπει να λάβουμε από την τελευταία κρίση και σε σύγκριση με το κράχα της δεκαετίας του 30 καθώς επίσης και το ποια πρέπει να είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία για το μέλλον. Να πω ότι επί της αρχής έχουμε μια στρατηγική η οποία θα έπρεπε να λειτουργήσει καλά και κατά τη γνώμη μου λειτουργήσε καλά έχουμε μεσοπρόθεσμους προσανατολισμούς για την δημοσιονομική πολιτική που μας δίνουν τη δυνατότητα για ελιγμούς επίσης και αν έχουμε πλεονάσματα εγκαίρως κάτι που βεβαίως δεν ήταν εύκολο να γίνει στις περισσότερες χώρες αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα όπως επίσης υπάρχει και καλή πολιτική παρακολούθησης. Άρα αυτό που πρέπει να τονίσουμε στα διεθνή φόρα είναι ότι υπάρχει προσέγγιση και υπάρχει προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι η κρίση δεν ξεκίνησε στην Ευρώπη, ξεκίνησε αλλού. Αλλά είχαμε ως Ευρώπη σημαντικές συνέπειες και τώρα που προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια παγκόσμια στρατηγική για την πρόληψη ή την μείωση των επιπτώσεων τέτοιου είδους κρίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν μεσοπρόθεσμοι προσανατολισμοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν Επίσης, για εμένα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο χαμηλός πληθωρισμός και η σταθερότητα των τιμών είναι προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη και θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, έχω κάνει και εγώ αλλά και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, για το θέμα δημοσίως. Εγώ σχολίωσα μόνο ένα σημείο κάποια στιγμή χωρίς να γνωρίζω όλα τα στοιχεία της παρουσίασης ε, του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών για αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Από τότε έχουν προκύψει και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Αφορά θέματα ελέγχου παρακολούθησης, κυρώσεων, προσφορά στήριξη, αλλά επίση έχουν συμπεριληφθεί πλέον και άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, επιτρέπουμε μία κήρυξη πτώχευσης από χώρα επιτρέπουμε έξοδο από την ευρώ Αυτά είναι θέμα που πρέπει να τα δούμε υπό την κατάλληλη προοπτική και να τα εξετάσουμε λεπτομερώς. Επίσης έχει ήδη τεθεί το ερώτημα αν θα χρειαστεί αναθεώρηση των συνθήκων. Όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020, είναι σημαντικό, όπως υπόθηκε και πριν, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για αύξηση της παραγωγικότητας. Η στρατηγική για το 2020 προσανασολίζεται στον, στην παραγωγή στο τέλος της οικονομικής δραστηριότητας δηλαδή. Όταν μιλάμε για παραγωγικότητα, μιλάμε για παραγωγικότητα και της εργασίας και σε αγαθά. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, κάτι που ήδη έχει υποθεί βεβαίως. Και το σημαντικό είναι το πώς θα μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της οικονομίας. Θα το μετρήσουμε με βάση τις εκροές της οικονομικής διαδικασίας. Χωρίς να μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, αν θέλετε, όσον αφορά τους προϋπολογισμούς. Υπερβολικές δαπάνες και μικρά έσοδα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό το θέμα τέθηκε το ερώτημα τι εισοδήματα χρειάζονται οι κυβερνήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Καταρχάς πρέπει να εξετάσουμε τις υποχρεώσεις. Είναι όλα όσα κάνουν οι κυβερνήσεις όντως ε, δημόσιες υποχρεώσεις του δημοσίου. βλέπουμε σε πολλές χώρες ποσοστά 80-90% του ΑΕΠ ως δημόσιο χρέος. Για να μειωθούν οι δαπάνες, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μία εξισορρόπηση και με τα έσοδα. Βεβαίως το ερώτημα που ετέθη ήταν ε, από πού θα προκύψει η ανάπτυξη και τι θα γίνει με την ε, κατανάλωση των ιδιωτών. Σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έμεση φόροι τα τελευταία δέκα χρόνια αυξάνοντας τους έμεσους ε, φόρους οι κυβερνήσει μείωσαν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όντως, Άρα πρέπει να εξετάσουμε και τις δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου. Όμως δεν μπορούμε να ξεκινάμε με σημείο εκκίνησης ότι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης πρέπει να μένουν αμετάβλητες. Πρέπει να δούμε με κριτική ματιά και αυτές τις υποχρεώσεις του δημοσίου. Όσον αφορά τις κυρώσεις, όντως δεν έχουν λειτουργήσει. Απέτυχαν το 2003 συγκεκριμένα και η συνέπεια ήταν ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης χρειάστηκε να αναθεωρηθεί προκειμένου να ενισχυθούν η δημοσιονομική κανόνες από τη μία πλευρά και από την άλλη να βρεθεί μια νέα διαδικασία για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Κάτι που δεν θα σημαίνει αλλαγή των συνθήκων, αλλά ίσως καλύτερη κατανόηση μεταξύ των υπουργών μεταξύ ειδικά των αμαρτωλών υπουργείων. Αν και βεβαίως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσει στους ενδυνάμει αμαρτωλούς. Έχουμε λοιπόν πολλούς δημοσιονομικούς κανόνες και πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι που δεν ισχύει σε άλλες περιοχές στον κόσμο και ευνοήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο που διαθέτει γιατί μας επιτρέπει μια συντονισμένη έξοδο από αυτό το πακέτο κινήτρων που χρησιμοποιήθηκε τώρα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι ο κύριος Στάρκμαν είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι θα έπρεπε να φύγει στις 5. Άκουσε όμως πολλές από τις παρουσιάσεις και τις ερωτήσεις που έχουν γίνει και βεβαίως ε, τώρα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και μεταξύ μας. Ο κύριος Κουσελάς από την Ελλάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος όλυρέν η Ελλάδα έχει πάρει όλα τα μέτρα, μέτρα επώδυνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, η επίθεση των κερδοσκόπων συνεχίζεται. Και δεν είναι επίθεση που αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι επίθεση που αφορά την Ευρωζώνη, είναι επίθεση που αφορά το ίδιο το ευρώ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν έχετε αποφασίσει για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των κερδοσκόπων και για την θωράκιση της Ευρωζώνης όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον από παρόμοιες επιθέσεις. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι ότι επειδή είναι δεδομένο ότι ο οικονομικός κύκλος εξόδου από την κρίση δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες, εάν κυρία Πρόεδρε θεωρείται ρεαλιστικό να γίνει προσαρμογή των κριτηρίων αποδοχής των ομολόγων που λαμβάνονται σαν εγγύηση για τη χρηματοδότηση κάθε χώρας ανάλογα με το πρόγραμμα σταθερότητας που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα. Και τέλος πιστεύετε ότι πρέπει σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που διανύουμε να απαγορευτεί η αγορά των CDS από ιδρύματα ή επενδυτές που δεν κατέχουν, δεν έχουν στα χέρια τους αντίστοιχες ομολογίες. Και μία τελευταία ερώτηση η κρίση την οποία περνάμε συνολικότερα όλες οι χώρες έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην απασχόληση με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Πιστεύετε ότι θα πρέπει η ανάπτυξη για την οποία μιλάμε να συνδεθεί με την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και με την προστασία ήδη υφιστάμενων θέσεων και αν ναι, με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση της ανάπτυξης με την απασχόληση για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. I'm Διαρωτώ με κατά πόσο θα απαντήσετε εσείς τώρα, κύριε Στάρκ, στο ζήτημα της κερδοσκοπίας και των CDS προτού να αποχωρήσετε. Πολύ σύντομα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση για το 2010 ανέλαβε μέτρα και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η εφαρμογή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντυπωσιάστηκε από αυτό το βήμα προς τα εμπρός και γνωρίζουμε ότι και η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο γνωρίζει ότι αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Πάντως σε κάποιες χώρες η διαδικασία θα κρατήσει πολλά χρόνια προκειμένου να μειωθεί και το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος και να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη πορεία. Τώρα, θα πρέπει να συζητηθεί και συζητάτε σε πολιτικό επίπεδο το θέμα των CDS. Σίγουρα Είμαστε πολύ διστακτικοί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις χρήσεις και συζητάμε πολλά θέματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο η κατάργησή τους, η απαγόρευσή τους θα ήταν η κατάλληλη λύση. Σίγουρα όμως χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και βελτίωση των υποδομών της αγοράς. Όσον αφορά τώρα την κερδοσκοπία, σίγουρα υπάρχει η κερδοσκοπία αυτή τη στιγμή, όμως είναι δύσκολο εξαιρετικά να την ποσοτικοποιήσουμε. Άρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τους κερδοσκόπους είναι να αποκτήσουμε αξιόπιστη πολιτική και αυτό έκαναν η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ίσως θα έπρεπε να πω στον ε, Έλληνα συνάδελφο ότι είχαμε το πρωί μία ακρόαση για τα παράγωγα και πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία. Μας επισκέφθηκε και ο Γκάρι Γκάνσλερ, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος ε, στην Αμερική για θέματα στην Επιτροπή για τα αμοιβαία και άλλα προϊόντα και συζητήσαμε το θέμα των ε, γυμνών παραγόντων και το κατά πόσο θα έπρεπε να απαγορευθούν. Αυτός όμως είναι υπέρ του να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση οι ελεγκτικές αρχές και να επιβάλλουν περιορισμούς στις θέσεις στον όγκο των συναλλαγών. Αυτά είναι πράγματα βεβαίως που θα συζητηθούν στο μέλλον και προετοιμάζει και η Επιτροπή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία έκθεση για το θέμα. Με συγχωρείτε που απαντώ εδώ εγώ, αλλά επειδή είχαμε την ακρόαση το πρωί, σίγουρα αυτό δεν αντανακλά τις απόψεις όλων μας, αλλά αποτελεί μια σύντομη σύνοψη. Ο κύριος Σίπ από την Γερμανία. Ja, Ευχαριστώ. Αν δούμε την στρατηγική του 2020 ως έχει, θα πρέπει να αναρωτηθούμε μετά από αποτυχίες ε, ξεκινάμε έναν ε, δρόμο που μπορεί να μας οδηγήσει πάλι σε κρίση. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι η όλη διαδικασία σχετικά με τον προβληματισμό και για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ε, απαιτεί μια περαιτέρω εμβάθυνση. Είναι... Μέχρι τώρα είχαμε ένα μια μορφή ανάπτυξης ε, που στηρίχθηκε στην, ε, στον δανεισμό τόσο σε ό,τι φορά τα κράτη όσο και τους ιδιώτες. Υπήρξαν κράτη τα οποία όμως μπόρεσαν να υποφελθούν από την κατάσταση. Πάρουν παράδειγμα τη Γερμανία. Το 1 τρίτο των εξαγωγών μας ε, κατευθύνεται προς χώρες οι οποίες σήμερα έχουν την περίφημη αυτή ονομασία PIGS το γερμανικό ΑΕΠ θα ήταν διαφορετικά πολύ χαμηλότερο. Και τώρα είναι αναγκαίο, πιστεύω, μια άλλη ατραπός να ακολουθηθεί για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι προσανατολισμός μας. Κάποιος, κάποιες παλές ιδέες που κατοχυρώνονται για παράδειγμα στη Γερμανία με ένα ωραίο νομοθέτημα που αφορά την ισορροπία όσον αφορά το εξωτερικό, τα, τις εξωτερικές μας εμπορικές σχέσεις που πρέπει να επανεξεταστούν, να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Είναι χρήσιμο αυτό στο οικονομικό αδιέξοδο. Αντί τα κονδύλια αυτά για να, να διατίθενται στην έρευνα και ανάπτυξη, να διατίθενται στις τράπεζες. Θα πρέπει τώρα αναπτυξιακά να δραστηριοποιηθούν δραστηριοποιηθούμε προς ε, μια σωστή πορεία και θα πρέπει να είναι τα κείμενα πιο φιλόδοξα ώστε να επιτευχθεί μια εκβάθρον αναθεώρηση του οικονομικού προτύπου και να προαχθεί ο στόχος αυτός και αυτά τα πρότυπα. Δεύτερο σημείο Πιστεύω ότι όσον αφορά τα όσα αναφέρθηκαν από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου όσον αφορά την οικονομική διαχείριση είναι κάτι που πολύ σοβαρά πρέπει να λάβουμε υπόψη διότι αυτό πιθανώς και στην αστοχία, στη μη επίτευξη του στόχου στο παρελθόν με την ατζέντα που είχαμε θέσει αυτό συσχετίζεται με το ότι τα μέσα που χρησιμοποιήσαμε δεν ήταν τα πιο ενδεδειγμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και τρίτον θα πρέπει, αυτή είναι η τελευταία παρατήρηση, να ξανασυζητήσουμε να δούμε αν οι διαφορετικές διαρθρώσεις και μηχανισμοί που έχουμε στα χέρια μας οδηγούν σε μια συνεπή πολιτική. Αν δηλαδή ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα μας οδηγήσει προς την κατεύθυνση που να ταιριάζει με αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αν όλα αυτά ταιριάζουν με τις οικονομικού τους οικονομικούς προσανατολισμούς που έχουμε ενώπιον μας. Αν σκεφτούμε ότι όσον αφορά το 2011 δεν μπορούν αυτά τα κίνητρα να ε, πάψουν ξαφνικά να λειτουργούν και τώρα Πολλά κράτη θέλουν ξαφνικά να εξοικονομήσουν κονδύλια και να έχουν περικοπέ. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτό θέτει το θέμα τη συμβατότητα και συνεκτικότητα τη πολιτική στην Ευρώπη. Και αν αυτό συσχετίζεται με το ότι δεν πετυχαίνουμε πολλού στόχου, οικονομικού στόχου, διότι δηλαδή δεν είναι συμβατή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Κίπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφό μου, ο Γκέρτ, είπε μέρο αυτών που θα ήθελα εγώ να πω Μπορώ λοιπόν έτσι να είμαι πιο σύντομος εγώ, όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ο ίδιος ότι μάλλον και για να το εκφράσω αήπια κάπως με για την απουσία ευρωπαϊκού πνεύματος και αξιών και αρχών σε όσα αναφέρθηκαν σήμερα εδώ. Όχι μόνο από τους δύο ε, εκπροσώπους που παρενέβησαν που δεν ε, είναι πλέον παρόντα, παρόντες, αλλά αν δούμε την πολιτική και τους στόχους μέχρι το 2020 και το ότι ούτε καν αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων, παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τη συνθήκη Λισαβόνας, υπό το άρθρο 121 εδάφιο 6, έχει περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά την οικονομική οικονομική πολιτική και τη χάραξή της κάτι παραπάνω από με εκπλήσει πρέπει να πω αυτό. Δεύτερο, θα έλεγα ότι αν και πάλι ξαναδούμε τη συνθήκη και τους βασικούς στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκρίνουμε όλα αυτά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, βλέπω μεγάλες διαφορές. Υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα να περιορίσουμε τις ανισότητες. Κάνουμε λόγο για την οικονομία, την κοινωνική οικονομία της αγοράς που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην αηφορία της ανάπτυξης ε, ως αρχές. Όμως, όσα παρουσιάζονται ως στρατηγική μέχρι το 2020 και οι δείκτες αυτής της στρατηγικής, τότε εξαχνίζεται, εξαερώνεται η ε, κοινωνική αυτή πολιτική και με το να ανταποκριθούμε στα λόγια μόνο, στη διατύπωση, ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες ε, της οικουμένης. Όλα αυτά δεν επαρκούν στο να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων και να, αναχαιτιστεί κλιματική, να οι κλιματικές αλλαγές. Αν δεν λάβουμε υπόψη την αποτελεσματικότητα της ε, χρήσης των πόρων, ε, των πρώτων υλών και την συμβατότητα με τους στόχους, αυτά τα οποία είχαμε πριν από 10 χρόνια όταν ξεκίνησε τη συνθήκη της Λισαβόνας, αν αυτά τα είχαμε πάρει στα σοβαρά, τότε <clears throat> δεν θα είχαμε φτάσει σε ένα διέξοδο φτάσαμε σε ένα διέξοδο με αυξημένους δείκτες όσον αφορά την χρήση των ε, ε, πρώτων υλών και τις ε, εκπομπές ρήπων. Υπάρχει εδώ κάτι που ούτε καν αναφέρθηκα, αναφέρθηκε από τους ομιλητές. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν είναι στο πνεύμα των συνθήκων, δεν, είναι, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της αλληλεγγύης, ούτε ανταποκρίνεται στο πνεύμα του, του, το ευρωπαϊκό. Και τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να αναφέρω το ίδιο, το ίδιο ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο θα υπομειστεί το κόστο τη προσαρμογή λόγω των ανισοτήτων που είναι τόσο οξυμένε, τόσο έντονε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το πώ εγώ κατανοώ τη διεθνή οικονομική κατάσταση και όσον αφορά και την κατανόησή μου των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπεριλαμβάνουν την αλληλεγγύη, το κόστο αυτό δεν μπορεί να το επομισθούν ε, οι χώρε ε, που ε, πιέζονται ιδιαίτερα και είναι αναπτυσσόμενε χώρε. Εδώ τέθηκε αυτό από τον Επίτροπο ε, Ρεν, ότι οι χώρες με ελλείμματα πρέπει να υπομισθούν, λέει, αυτό το βάρος. Δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο ούτε και από τους ε, ε όσους εκπροσωπούν τις χώρες με πλεονάσματα. Όμως ε, για να λειτουργήσει κάτι, για να χορέψει κανείς χρειάζεται έναν παρτενέρ, έναν εταίρο. Αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πράγματα. Διαφορετικά το επίπεδο του ε, κόστους προσαρμογής το οποίο θα επομισθούν οι χώρες με ελλείμματα θα είναι ανέφικτο και οικονομικά και πολιτικά. Δεν νομίζω να είμαστε αρκετά σοβαροί εδώ για τους πραγματικούς κινδύνους ε, να υπάρξει κατακαιρματισμός ή διχασμός ε, της διαδικασίας ολοκλήρωσης λόγω του επίπεδου στο οποίο έχουμε φτάσει. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και κανόνες όπως έχουν εκφραστεί από τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα επανέλθω. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Στάρκα διότι παρατείνει την ε, παραμονή του ανάμεσά μας όσο γίνεται περισσότερο για να μπορεί και αυτός να συμμετάσχει και να αντιδράσει. Μάλιστα σωστό για τις δύο τελευταίες αυτές παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις. Πρώτα, εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική για τη Λισαβόνα δεν απέτυχε. Όχι κύριοι. Εντάξει, μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση και μετά την επικέντρωση για το ότι η στόχη ήταν πιο στοχοθετημένοι, πιο σωστά μετρημένη. Η Λισαβόνα, η συνθήκη τη Λισαβόνα έδωσε θετικά αποτελέσματα. Όμω η κρίση κατέστρεψε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να πούμε. Η κρίση κατέστρεψε, υπονόμευσε αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ άλλων από, συνθήκη, από τη στρατηγική της Λισαβόνας δεν ήταν πλέον αηφόρα, δεν μπορούσαν να διατηρηθούν. Τώρα που έχουμε τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, το 2020 με επικέντρωση σε λιγότερους στόχους από ότι αρχικά με τη στρατηγική της Λισαβόνα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων, αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν πιστεύω, δεν βλέπω ότι πρόκειται για αδιέξοδο οικονομικά εδώ κύριε, όταν πρόκειται για τις ανισότητες, τις εσωτερικές ανισότητες στην Ευρωζώνη, σωστό, εντάξει, υπάρχουν χώρες ελληματικές και χώρες με πλεονάσματα. Όμως από την άλλη πλευρά, εσείς επιχειρηματολογείτε και λέτε ότι εκείνοι που παράγουν υψηλότερο επίπεδο χρέους θέτουν ακριβώς υψη, μεγαλύτερα εμπόδια και για τις χώρες που έχουν πλεονάσματα. Και εδώ πάλι όμως πιστεύω ότι κάποιες χώρες στη ζώνη ευρώ αλλά νομίζω μπορούμε να το πούμε και αυτό συνολικά. Κάποιες προηγμένες οικονομίες ζούσαν και δαπανούσαν περισσότερο από όσο μπορούσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ως περίπτωση εδώ, στη ζώνη ευρώ με ανάπτυξη ΑΕΠ κατά μέσο όρο περίπου 4%, σαφώς πάνω από τον όρο, μέσο όρο ανάπτυξη στη ζώνη ευρώ. Ταυτόχρονα με οξυμένη αύξηση των μισθών στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα σαφώς πάνω από το κέρδος στην αύξηση παραγωγικότητας βλέπουμε ότι όλα αυτά τα κόστη εξεράγησαν και η οικονομία αυτής της χώρας έγινε, ε, κατέστη, κατέστη λιγότερο ανταγωνιστική. Τι είναι λοιπόν το benchmark, το benchmark ε, το, ο μέσος όρος από πλευράς πλεονασματικών χωρών και ελληματικών χωρών. Ποια πολιτική, ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθηθεί το benchmark είναι σαφές. Δεν πρέπει να αποδυναμωθεί αυτό που επετεύχθη σε σχέση με χώρες που προσαρμόστηκαν αποτελεσματικά. Και το κόστος προσαρμογής πιστεύω εγώ τώρα, όπως είπε η Επιτροπή, είναι περισσότερο, περισσότερο πλέον θα πρέπει να το επομισθούν οι χώρες με ελλείμματα. Διότι ακριβώς αν δεν αλλάξουν τις πολιτικές τους θα συντριβούν. Είναι απλό. Και πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν όπως είναι αναγκαίο. Και ξέρουμε ότι μετά από ένα boom, μετά από μια ε, έκρηξη ανάπτυξης, υπάρχει ανάγκη, μεγάλη ανάγκη αναδιαρθρώσεων και προσαρμογών και αλλαγή στην πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτό κάνουν τώρα οι χώρες αυτές, αυτό που έκανε η Ιρλανδία και εξακολουθεί να πράττει. Και πρέπει να πω ότι η Ιρλανδία έλαβε πολύ γενναίες αποφάσεις και το ίδιο αληθεύει τώρα για την Ελλάδα. Η προσαρμογή λοιπόν είναι υπόθεση κυρίως των χωρών μελήματα. Και πάλι εδώ όταν έχουμε το θέμα προτύπου ανάπτυξης στο παρελθόν αλλά και για το μέλλον, εγώ θέλω να κάνω μια σαφή διαφοροποίηση. Αν αυτό το πρότυπο ανάπτυξης ε, έχει ως πρότυπο την αγορά ή την πολιτική policy driven. Υπάρχει μια πολιτική όσον αφορά στοχοθέτηση και στρατηγική για εξαγωγέ. Στρατηγική για εξαγωγέ που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ή οφείλεται σε μια αποκεντρωμένη διαδικασία και για μένα αποκεντρωμένη διαδικασία μπορεί να πει κανείς εντάξει ωραία θα ανταγωνιστείτε με άλλες χώρες, θα ανταγωνιστείτε παγκόσμια. Ε, τότε πρέπει λοιπόν να καταλήξετε σε διαφορετική κρίση, διαφορετική στάθμιση και να έχετε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρόεδρος ευχαριστώ. Κύριε Πισανή, θέλετε να απαντήσετε σύντομα εσείς, παρακαλώ. Okay, maybe, maybe on the same, the same ε, Επειδή τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, να πω ότι χρειάζεται να γνωρίσουμε πως ε, δεν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για να αποφασίζουμε σε ζητήματα όπως αφορά τα ισοζύγια πληρωμών. Αυτό είναι ζήτημα εντελώ διαφορετικό από το θέμα του προπολογισμού. Στου ε, προπολογισμού μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το χιέλημα, το χιπλαιόνασμα κλπ. Σε ό,τι αφορά όμω ε, τώρα τα ισοζύγιο ε, πληρωμών πρόκειται για αποταμιεύσεις οι οποίες πάνε από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια κρίση, μια απόφαση σχετικά το τι είναι καλό, τι όχι. Συνήθως τα, τα χρήματα πηγαίνουν από τις ε, φτωχές πλούσιες χώρες ε, αλλά και από τις πλούς φτωχές. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση είναι πολύ καλύτερο. Καλύτερα να βλέπουμε λοιπόν αποταμιεύσει από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε αποταμιεύσει να πηγαίνουν από τις πλούσιες τι ε, φτωχές. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, αυτό σημαίνει σύγκληση. Αυτό όμως είναι εντελώ διαφορετικό από το φορολογικό έλλειμμα. Και συνδέονται ελάχιστα στον παραδοσιακό τρόπο σκέψης για τους ε, στόχους της πολιτικής, της η φορολογική πολιτική σας οδηγούσε στο να επιθυμείτε να μην έχετε μεγάλα ελλείμματα αλλά και να φροντίζετε να υπάρχει Αλλά η κρίση τι έδειξε. Κατέδειξε ότι αυτό δεν συμβαίνει και η πηγή της ε, αστάθειας δεν προέρχεται μόνο από μια φορολογική ε, ένα φορολογικό πρόβλημα. Φυσικά προέρχεται και από κάτι τέτοιο για την, Ελλάδα, αλλά ρίχτε και στην Ισπανία μια ματιά να δείτε. Διότι οι δύο κρίσεις δεν προέρχονται από τον αυτό τρόπο και διαχείριση της οικονομίας. Αυτή λοιπόν είναι μια πνευματική άσκηση που θα πρέπει να μας απασχολήσει τα προσεχείς μήνες και έτη. Τώρα για να καταστώ πιο συγκεκριμένος το θέμα ότι χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς ταγκό. Να πω ότι οι χώρες με έλλειμμα θα μπορούσαν να αποτανθούν στη Γερμανία και να πούν γιατί εσείς έχετε πλεόνασμα. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και ε, αυθόρμητα μια ρύθμιση θα, δεν θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια τέτοια εξισορρόπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε πως στην παγκόσμια οικονομία η ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερη από αυτήν των ΗΠΑ. Τώρα, η Γερμανία έχει ένα πλεόνασμα, αυτό είναι πρόβλημα για μας, θα μπορούσαμε να πούμε, κάντε κάτι. Το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα ατομικής συμπεριφοράς και το άθροισμα αυτών των συμπεριφορών. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο γερμανικό πλεόνασμα και το κινέζικο πλεόνασμα. Πίσω από το κινέζικο πλεόνασμα μπορείτε να πείτε ότι υπάρχουν προφανείς στρεβλώσεις. Υπάρχουν στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση των ε, αποταμιεύσεων, σε ό,τι αφορά την ισοτιμία, την ανταγωνιστικότητα. Μπορούμε λοιπόν εν μέρη να πούμε ότι το πλεόνασμα οφείλεται σε κάποιες τρευλώσεις. Στην περίπτωση της Γερμανίας όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στην ε, Γερμανία το ότι υπάρχει το πλεόνασμα οφείλεται ενδεχόμενα και στο ζήτημα της συμβίωσης των μισθών είναι και αυτή μια αιτία. Η εξέλιξη σε θέματα υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα θα πρέπει να τα βλέπουμε ως συμπτώματα των προβλημάτων. Αυτά τα αυτά, ε, έλλειμμα και πλεόνασμα μπορεί να μην αποτελούν πρόβλημα, αλλά πρόβλημα μπορεί να είναι αυτό που τα προκαλεί. Και όπως είπε ο Λιρέν, έχουμε νομική βάση αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να αποκτήσουμε είναι η ε, σκέψη για την εξέβρεση λύσης. Τώρα για την Λισαβόνα. Νομίζω πως η ε, Λισαβόνα είχε μια διάγνωση που εν μέρει ήταν ορθή. Γι' αυτό τη διάρκεια τη τελευταία δεκαετία Υπήρχε προβλήματα με τα ποσοστά απασχόλησης αλλά και με την καινοτομία. Υπήρξε μια αξιολόγηση η οποία ήταν σωστή. Αλλά υπήρχαν και κάποια στοιχεία που έλειπαν, όπως χάρη η εκπαίδευση. Υπήρξε εστίαση στην ανάπτυξη και την έρευνα, αλλά όχι στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Τώρα η πράσινη οικονομία σίγουρα δεν είχε τη θέση που απέκτησε σήμερα υπάρχουν κάποια στοιχεία που απουσιάζουν, όπως ε, τα χρηματοοικονομικά. Το θέμα της ε, ανάπτυξη ανάπτυξης και της σταθερότητας ε, και η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ανάπτυξη θα έπρεπε να έχει ένα πιο κεντρικό ρόλο στην όλη συζήτηση. Το ίδιο και τα δημοσιονομικά. Ε, έχουν, αποτελούν πλέον ένα κεντρικό ζήτημα. Κάτι που δεν υφιζόταν στο παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν τη σημασία που έχουν τα δημοσιονομικά στην οικονομία μας. Το, το θέμα των φόρων επίσης. Ποιοι φόροι θα πρέπει ή μπορούν να αυξηθούν και ποιοι όχι. Έχουμε πολλά λοιπόν να κάνουμε στον τομέα της φορολογικής πολιτικής. Τώρα για να ολοκληρώσω για τη διακυβέρνηση. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα ανίσχυρα εργαλεία σχετικά με το ότι θα πρέπει να γίνει και το ζήτημα της διακυβέρνησης μετά τη στρατηγική Λισαβόνας δεν έχει επιληθεί μέσω των νέων προτάσεων. Έχουν υπάρξει βελτιώσεις, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας είναι ικανά. Δέκα ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Προτείνω το εξή. Θα δώσω προτεραιότητα στα μέλη των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρώτα θα μιλήσουν να έρθει από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής ε, ΕΚΟ. Η κυρία Καλμάρη από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Φινλανδία υποστηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Ανησυχεί όμως η Φινλανδία ότι δεν θα πετύχει αυτή η στρατηγική. Εκτός αν, εκτός αν δεσμευτικοί όροι και προϋποθέσεις ως ορόσημα τεθούν κατά μήκος αυτής της πορείας και εκτός αν υπάρξουν κυρώσεις εις βάρος των χωρών που δεν θα είναι αποτελεσματικές και δεν θα συμμορφώνονται. Η παραγωγικότητα τώρα. Η παραγωγικότητα θα είναι όλο και πιο σημαντική, περισσότερο σημαντική από ό,τι οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και θα πρέπει μετρήσιμη να είναι, μετρήσιμη παραγωγικότητα. Και αυτό επειδή δεν μπορούμε να θυσιάσουμε το περιβάλλον, για παράδειγμα. Ε, όσον αφορά τον, έναν πιθανό ανταγωνισμό με τους Κινέζους. Το περιβάλλον δεν μπορεί να θυσιαστεί εις βάρος ενός τέτοιου ανταγωνισμού. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο οι ρυθμίσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η νομοθεσία θα διοργανώνεται παγκόσμια θα είναι ένα όλο και πιο σημαντικό στοιχείο. Ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με τα χρηματιστήρια όσον αφορά το MIFID. Δεν ξέρουμε όμως τι συμβαίνει εκτός χρηματιστηρίων. Αν θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των ε, εκτός θα έλεγα πλαισίου και κανονισμών συναλλαγών. Επίσης θετικό θα ήταν αν μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος παγκόσμια με την επίτευξη ενός φόρου ή τέλους στις παγκόσμιες συναλλαγές ως ένα είδος μέσου ώστε να μπορούν και οι συναλλασσόμενοι να συνεισφέρουν σε σχέση με αυτό το κόστος και τις δαπάνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μινάρη παρακαλώ πάλι από την Φιλανδία. Uh, uh, Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ πρώτον να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω λοιπόν για αυτήν την συνεδρίαση, για αυτήν την συνάντηση μαζί σας. Και να πω ότι προφανώς εδώ σε σχέση με την ε, γλώσσα μου θα ήθελα να συνεχίσω στα φινλανδικά. Λοιπόν, είναι σαφές ότι η μοίρα, το πεπρωμένο του ευρώ είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα. Για να το δούμε αυτό. Δυστυχώς ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απουσιάζει, αποχώρησε. Παρέμεινε μετέωρη η ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Πολλές χώρες έχουν ε, πραγματικά προσδοκούσαν την βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική αν μήπως μελλοντικά θα ήταν δυνατό να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ρυθμιστικά τώρα, εφόσον και καθώς υπάρχουν διεθνείς συναλλαγές ε, με ευρωπαϊκές τράπεζες, είπα, αμερικανικές τράπεζες εδώ και αλλού παγκόσμια, δεν παίζει ρόλο αν ε, διοργανώσουμε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν γίνει κάτι παρόμοιο στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου παγκόσμια. Δυστυχώς όμως κάποιες εκπλήξεις μπορούν να χτυπήσουν, να πλήξουν την Ευρώπη. Εκπλήξεις από γεγονότα ε, από το εξωτερικό, τον έξω. Και αυτό ζήσαμε στη Φινλανδία κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1990 και έπρεπε να πληρώσουμε τα σπασμένα εμείς οι ίδιοι. Ολοκληρώνοντα εν κατακλείδη, θα ήθελα να αναφέρω την συνεδρίαση, την σύνοδο της Κοπενχάγη. Ήμουν εκεί όταν απέτυχε να επιτύχει, να επιτύχει τους στόχους της αυτή η συμφωνία. Ο Σαρκοζή είπε ότι κατά τη διάρκεια δηλαδή όταν στις 12 η ώρα θα υπήρχε λέει συμφωνία, υπήρχε λέει συμφωνία. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα αναπτύξει την συνεργασία της η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν έχει ε, ιδιαίτερο βάρος και θα ήθελα να ξέρω πώς αυτό θα αποφευθεί στο μέλλον. Και μετά για τους δείκτες του ΑΕΠ είναι αξιόπιστοι δείκτες ε, για χώρες ε, και την ευημερία τους. Δεν θα έπρεπε να εξετάσουμε δείκτες όπως το δίκτυ δίκτυο για παράδειγμα, δίκτυ αθλητισμού, δίκτυ πολιτισμού και συναφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για αυτή την τελευταία παρατήρηση μπορώ να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια έκθεση που αναφέρεται ως σε τίτλο «Το ΑΕΠ και πέρα από το ΑΕΠ» και από κοινού και όλα και ε, με, τη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, έχουν αναλυφθεί δράσεις. Επόμενος, ο κύριος Τσούμβολς από την Αυστρία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, δεν θα θέσω ερωτήσεις, επειδή η πλειοψηφία έχει αποχωρήσει από τους εισηγητές. Θα ήθελα όμως να μεριμνήσετε μελλοντικά να διασφαλίζετε όταν πανευρωπαϊκά έχουν, έχετε βουλευτές εκπροσώπους εδώ ανάμεσά σας, για κάποιες λίγες ώρες οι εισηγητές να είναι παρόντες. Θα το παρακαλούσα θερμά για το μέλλον. Λοιπόν, μια σύντομη παρέμβαση από πλευρά μου χωρίς ερωτήσεις. Όλοι συμφωνούμε το 2010 είναι έτος κλειδί για μας. Αν δεν καταφέρουμε, αν δεν τα καταφέρουμε να πετύχουμε μια αηφορία όσον αφορά την ανάπτυξη και να την δρομολογήσουμε, απειλεί ο κίνδυνος τότε. Η Ευρώπη να καταλήξει σε μια θέση σάντουιτς μεταξύ της δυναμικής των ασιατικών χωρών αφενός και των ΙΠΑ αφετέρου. Και τώρα για τον ρόλο της στρατηγικής 2020. Πρέπει να προσθέσω την φωνή μου στους προλαλήσαντες που είπαν και πίστεψαν ότι σε πολλά ε, τους θύμισαν αυτά τα πράγματα την στρατηγική της Λισαβόνας. Θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο Στάρκ όταν λέμε ότι απέτυχε η στρατηγική λέει της Λισαβόνας μόνο και μόνο επειδή ξέσπασε η οικονομική κρίση. Αν δει κανείς τις ε, εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συγκρίνει με τις, αιτήσεις, εκθέσεις ε, προόδου της Business Europe τότε πολλά βρίσκονται ενδιάμεσα όταν λένε ότι για παράδειγμα η Business Business Europe είναι πολύ πιο επικριτική στις παρατηρήσεις. Από τις αδυναμίες της στρατηγικής ε, της Λισαβόνας πρέπει κάτι να μάθουμε και να μην λέμε ότι όλα πήγαν με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ υπάρχουν πολλά ευάλωτα σημεία. Πρώτον, όλοι μας πιθανότατα και πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ήταν λαμπροί όσον αφορά τη ρητορία τους και τους λόγους που εκφωνούσαν. Ήταν όμως υπερβολικά ευάλωτοι και αδύναμοι στις πράξεις. Αποτελεσματικός όμως είναι εκείνος που κάνει πράξεις. Πολύ λιγότερο λιγότερα γίνονται από τους ρήτορες και τους μεγαλώς, τις μεγαλόστομες διακηρύξεις. Όποιος πιστεύει ότι απλά και μόνο η θέσπιση φιλόδοξων στόχων είναι το σημαντικό στο έγγραφο για στρατική 2020 και ότι όλα αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα, να μπορούν να αναπτύσσονται, να υπάρχει διαρκής εποπτεία και επιτήρηση. Και όταν λέμε κυρώσεις, κυρώσεις στην πραγματική ρεαλιστική πολιτική δεν είναι εφικτές. Και όταν λέμε καλύτερα είναι τα κίνητρα και τα θετικά αντί τα αρνητικά και οι κυρώσεις, ε, τότε πρέπει να, πολλά να φανταστούμε για να πετύχει η πολιτική αυτή των κινήτρων. Διότι φοβάμαι κατά τα άλλα ότι αυτή η ίδια η στρατηγική μας θα έχει την ίδια μοίρα, την ίδια έκβαση όπως η προηγούμενη στρατηγική για τη Λισαβόνα. Αποτυχία δηλαδή. Λιγότερους στόχους να έχουμε, μετρήσιμους, με εποπτεία, τηρήσιμους. Αυτό θα ήταν για μένα πολύ σημαντικότερο από πολυάριθμους στόχους που δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Πέντε παραδείγματα. Σταθεροποίηση των οικονομικών αγορών. Δεύτερον, εξυγεία εξυγίανση των δημοσιονομικών με μεταρρυθμίσεις και διαθωτικές μεταβολές, αλλαγές, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγορές, έρευνα, ε, <clears throat> ανάπτυξη. Αν καταφέρναμε αυτούς τους πέντε στόχους να υλοποιήσουμε θα, είχαμε, θα ήταν επιτυχές το εγχείρημά μας. Ευχαριστώ. Κάπως ξεπεράσατε το χρόνο σας. Ο κύριος από την Αυστρία, ο δεύτερος ε, βουλευτής από την Αυστρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ άμεσα μπορώ να συνεχίσω μετά την παρέμβαση του προλαλήσαντος Γκούντερ. Όμως δύο ερωτήσεις θα ήθελα να διατυπώσω που ίσως ενδιαφέρουν τους ε, κυρίους ε, στο βήμα από την Αυστρία. Για μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι δύο τρίτα όλων των απασχολουμένων μας απασχολούν στην Αυστρία. Και είναι νομίζω και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, κάτι παρόμοιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η οικονομία είναι οι πιο αξιόπιστοι πυλώνες, ο πιο αξιόπιστος πυλώνας της οικονομίας κατά την δύσκολη περίοδο 2008-2009. Και κατά την διάρκεια της κρίσης τα κατάφεραν καλύτερα από τους άλλους όσον αφορά την απασχόληση. Γι' αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω Χρειαζόμαστε ρυθμιστικό πλαίσιο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ υπήρξε και υπάρχει ένα καλό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η α, απαλλαγή όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, και την επισκευή ε, ΙΧ αυτοκινήτων συνολικά και το θέμα των υπηρεσιών όσον αφορά τα, τα αυτοκίνητα. Ακριβώς για την, τις υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων κατά το επόμενο διάστημα θα εκπνεύσει η διάταξη. Και εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι εκ νέου θα είναι εξάρτημα ή αγόμενο, σειρώμενο, φερόμενο των μεγάλων βιομηχανιών. Πρέπει να μεριμνήσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατευτούν. Και θέλω ρητά και κατηγορηματικά να πω ότι αυτό είναι μείζον πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της επισκευής και παροχής υπηρεσιών για τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Σπότης από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, πέρα από τις στρατηγικές, τα προγράμματα και τις συζητήσεις, πρέπει να επικεντρωθούμε στους στόχους της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 9%, 30 εκατομμύρια άτομα. Και δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους που ενδεχομένως ήταν υπερβολικά φιλόδοξοι. Ούτε υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση της ε, οικονομικής σύγκλησης αυτή τη στιγμή για κάποιες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ποσοστό ρεκόρ ανεργίας ε, των ε, νέων κάτω των 25, 25% ανεργία τι είδους λύσεις μπορούμε να βρούμε για να εντάξουμε τους νέους στην αγορά εργασίας. Και επειδή έχουμε και πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες των νέων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι προτείνει η στρατηγική για το 2020 για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 35 ετών. Ευχαριστώ. Θα περάσω τώρα στους ευρωβουλευτές. Ε, υποθέτω ότι θα θέλετε και να απαντήσετε σε ορισμένες σχετικές ερωτήσεις. Το λόγο έχει πρώτα ο κύριος Τσικλούνα. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που σας βλέπω πιο επικριτικούς όσον αφορά κάποια συνθήματα όταν δεν ακούγονται όντως πιστικά. Και αυτό το ακούω και από τους εθνικούς, ευρωβουλευ... Ε, και από τους εθνικούς βουλευτές και από τους ευρωβουλευτές. Βλέπουμε μία στρατηγική σαν να είναι ένα μοντέλο που μπορούμε να ακολουθήσουμε οδηγίες από κάποιο βιβλίο, ενώ δεν υπάρχει τέτοιου είδους προσέγγιση. Μας λέτε ότι ο ένας πυλώνας είναι η εξυγίανση και ο άλλος η ανάπτυξη. Αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ελληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε ενθουσιασμό για αυτή τη στρατηγική για το 2020 όταν αυτή τη στιγμή το μόνο που σκεφτόμαστε είναι μία λέξη. Χρέος. Δημόσιο χρέος. Ναι, είναι σαν να βρισκόμαστε σε κούρσα και χρειαζόμαστε στόχους, στρατηγικές, ανθρώπινους πόρους, τεχνολογία. Όμως, από την άλλη πλευρά, βρισκόμαστε σε μία βάρκα που έχει τρύπα και μπάζει νερά, ενώ πρέπει να συμμετέχει σε κούρσα. Άρα, ακόμη και ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε για τις επιδιορθώσεις, τις επισκευές, είναι καλά αξιοποιημένος. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να είναι απόλυτα λογική γιατί το μυαλό τους έχει σκοτεινιάσει από τα όλα όσα ακούνε για την κρίση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι κυρία Ποδηματά, παρακαλώ. Um, Ο κύριος Όλε Σμιτ λοιπόν τότε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη ευκαιρία αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Όχι μόνο με τα μέλη στο πάνελ αλλά και με τους άλλους συναδέλφους. Είμαι ευρωβουλευτής από τη Σουηδία και είμαι φιλελεύθερος. Αυτά σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία για το άτομο μου. Πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη ήταν διχασμένη. 15 χρόνια είχαμε πολέμους στα Βαλκάνια. Δεν νομίζετε ότι είμαστε καλύτερα τώρα πια. Και κατά τη διάρκεια του 1930 μια παρόμοια κρίση είχαμε. Όλοι ξέρετε που κατέληξε. Κατέληξε σε προστατευτισμό. Κυρίως ο προστατευτισμός που παρέμεινε εκτός σε αυτή την κρίση τώρα. Λοιπόν, να μην βλέπουμε πάντα τη μαύρη τρύπα και τα αρνητικά και να λέμε ότι όλα είναι ανέφικτα, αδύνατα και αρνητικά και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Δεν θα πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Αλλά ούτε και υπεραπεσιόδοξοι διότι η απεσιοδοξία αυξάνεται, μεγαλώνει και φτάνει πια αυτό, αρκετά το ζήσαμε. Ένα σχόλιο όσον αφορά τους Έλληνες συναδέλφους. Νομίζω όλοι μας εδώ σε αυτή την αίθουσα σας υποστηρίζουμε. Γνωρίζουμε το τι κάνετε. Και αυτό που κάνει το έργο σας είναι πάρα πολύ άκρος δύσκολο. Βρισκόμουν στη θέση σας, βρισκόμαστε στη θέση σας ε, τη δεκαετία του 1990, ε, κατά τη διάρκεια της ε, δεκαετίας του 1990 στη Σουηδία. Είχαμε τεράστια ποσοστά επιτοκίων και τα λοιπά και είχαμε αποτυχία και είχαμε και εμείς κερδοσκόπους. Ο κύριος Τζόρτζο Σόρος ήταν ο κύριος κερδοσκόπος όσον αφορά και τον, ε, την κερδοσκοπία με την ε, ε, στερλίνα λίρα, στερλίνα της Αγγλίας και την κορώνα της Σουηδίας. Δεν θα πρέπει να πυροβολεί όμως κανείς τον πιανίστα. Εσείς κάνετε προσπάθειες, αλλά μην, επικεντρωνόμαστε, μην επικεντρώνεστε υπερβολικά στους κερδοσκόπους. Αυτό χρησιμοποιείται υπερβολικά νομίζω θα έλεγα εγώ. Θα, σε ευχόμουν καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας ολόθερμα. Κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας, εγώ προέρχομαι από μια σκανδιναβική χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία που προσπαθούσατε να πετύχετε με την Ισλανδία όσον αφορά το Ice Save, νομίζετε ότι είναι αξιοπρεπή συμφωνία αυτή. 50.000 άνθρωποι που προσπάθησαν να εκταμιεύσουν και να διασώσουν ό,τι ήταν δυνατόν από τράπεζες κτλ. Δέχεστε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή του iSave. Είναι αξιοπρεπής. Νομίζω είναι τελείως αναξιοπρεπής και από πλευράς κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και από πλευράς κυβέρνησης Ολλανδίας. Εγώ θα ήθελα σε σχέση με το τελευταίο να δούμε, αλλά υπάρχει κάποιος από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία που θα ήθελα να απαντήσει. Δεν βλέπω κανένα να σηκώνει το χέρι του. Α, εσεί, ωραία, πολύ σωστά. Από την Ολλανδία θα έλεγα. Εσεί, λοιπόν έχετε τον λόγο. Μέβε το όνομά μου από την ε, Ολλανδία και εγώ φιλελεύθερο είμαι. Και αισθανόμαστε ότι ευελπιστούμε και έχουμε εμπιστοσύνη. Είμαστε πισμένοι ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Μια τέτοια συμφωνία δηλαδή με τους Ισλανδούς. Με την κυβέρνηση της Ισλανδίας λοιπόν. Ευχαριστώ. So are we. Εντάξει και αν βλέπω καλά η Βαρόνι Κόεν. Φοβούμαι συμφωνώ πρέπει να πω με τον Ολλανδό συνάδελφο επ' αυτού. Γνωρίζετε έπρεπε να πληρωθούν ε, δικοί μας πολίτες και αισθανόμαστε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να πληρωθούν ε, από πλευρά των Ισλανδών να καλυφθούν. Ευχαριστώ. Um, Ωραία, εντάξει. Θα έλεγα εγώ ίδια ίσως θα έλεγα ότι υπάρχει δικαίωμα ανάκτησης κονδυλίων, αναπλήρωσης κονδυλίων, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά ε, πολύ τιμωρητικά επιτόκια όσον αφορά ε, την ε, αποπληρωμή αυτών των ποσών. Κάτι θα έπρεπε να γίνει να είναι πιο δίκαια, πιο ισοδίκαια η κατάσταση. Για να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Πόρτας, θέλατε εσείς να επανέλθετε, ίσως σύντομα όμως παρακαλώ και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Πιζανή να δώσει τις τελικές του παρατηρήσεις. Κύριε Πόρτας, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ ομολογώ ότι αν ήμουν Ισλανδός και εγώ θα είχα τις δικές μου αμφιβολίες στο να δοθούν περισσότερα δικαιώματα, περισσότερε περισσότερες ευκαιρίες όσον αφορά την κάτω χώρε τις κάτω χώρες και την, το Ηνωμένο Βασίλειο για μια πληρωμή, για μια χρήση, κρίση για την οποία δεν ήταν υπεύθυνοι οι ίδιοι Ισλανδοί. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στο πρόβλημα των μεγάλων ανισοτήτων στη ζώνη ευρώ. Και αυτό επειδή Πιστεύω ότι υπάρχει μια δυσκολία με το ευρώ. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Πιζανή. Και ουσιαστικά είναι το εξή. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν δυνατόν να αντέξουμε ένα νόμισμα που δρά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για χώρες που είναι έντονα ελληματικές στο εξωτερικό του εμπόριο ή για χώρες που είναι υπερβολικά πλέον ασματικές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό τι λέει. Πρόκειται για μια κατάσταση πολύ περίπλοκη που δημιουργείται, γιατί υποχρεώνει τις χώρες με ελλείμματα να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους και ακόμα να υποτιμούν κιόλα όλου του συντελεστέ παραγωγής, παραγωγικότητας γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συναλλαγματικέ ισοτιμίες για να είναι προ όφελό του. Αυτό που προηγούμενα γινόταν με υποβάθμιση, υποτίμηση νομίσματο, τώρα γίνεται με την υποτίμηση του κόστου παραγωγή, και ιδιαίτερα με υποβαθμίσει και υποτιμήσει των μισθών, μειώσει των μισθών. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ολόκληρη σειρά χωρών που ζουν εδώ με αυξήσει μισθολογικέ πάνω από την παραγωγικότητα παραγωγικότητά Εγώ είμαι Πορτογάλος. Αυτό που αυξήθηκε πάνω από την παραγωγικότητα ήταν το θέμα των πιστώσεων. Όχι οι μισθοί. Οι μισθοί έχασαν αγοραστική δύναμη κατά τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και γι' αυτό εδώ τίθεται, το εξής, τίθενται τα εξή ερωτήματα. Τα προγράμματα σταθεροποίησης τα οποία εξετάζονται και υλοποιούνται είναι προγράμματα τα οποία αναζητούν μια διέξοδο από την κρίση μέσω εμβάθυνσης της ίδιας της ύφεσης όμως. Θα έλεγα ότι η μόνη διέξοδος που βλέπω και είναι προφανής για την κρίση στην Ευρώπη και τη ζώνη ευρώ είναι να ζητήσουμε από τους Γερμανούς να αγοράζουν περισσότερα, να καταναλώνουν περισσότερα. Δηλαδή να υπάρξουν αυξήσει ε, μισθολογικέ που θα του δώσουν τη δυνατότητα να ζητούν να αγοράσουν περισσότερα και να αυξηθεί η αγοραστική του δύναμη. Και αυτό θέτει το τελικό ερώτημα με τον εξή τρόπο. Εμεί χρειαζόμαστε στη ζώνη ευρώ συντονισμό των πολιτικών μα. Χωρί καμιά αμφιβολία αυτό. Όμω, γιατί αυτό ο συντονισμό μα λέει ότι μέχρι το 2013 λέει θα γίνεται και όχι μέχρι το 2014 ή όχι μέχρι το 2015. Γιατί αυτό. Γιατί πρέπει έτσι να επιτευχθούν τα 3% του ε, ελλείμματος ε, και το 60% του χρέους. Και γιατί είναι 3% και όχι 5% ή παραπάνω. Όταν στις είπα το ε, έλλειμμα είναι 12%. Και γιατί το, να είναι το δημοσιονομικό χρέος 60% και όχι 90% του ΑΕΠ. Για παράδειγμα όσον αφορά το χρέος. Αν γίνει με συντονισμένο τρόπο. Γιατί λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Right. And, Sven, you had a final quick question. Sven, είχατε εσείς μια σύντομη τελική ερώτηση. Just would like to briefly... Εν να απαντήσω σε κάποια από τα επιχειρήματά σας και γιατί ανησυχώ τόσο για το επίπεδο των ανισορροπιών που η Ευρωζώνη αλλά και η Ευρώπη γενικότερα αντιμετωπίζει. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχουμε κάποια ελλείμματα τα οποία είναι δύνατον να διατηρηθούν και σε κάποιες χώρες έχουν φτάσει σε σημείο το οποίο δεν μπορούν με τίποτα να υπερβούν και εδώ διαφωνώ με τον συνάδελφο μου τον Πέτερς ε, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις ε, ανισότητες αυτές που υπάρχουν και είπατε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα νόμισμα σε μια περιοχή νομίσματος γιατί θα πρέπει να ανησυχούμε. Μα νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Αλλά θεωρώ πως δεν βρισκόμαστε σε μια ολοκληρωμένη ενία αγορά. Οι Έλληνες δεν μπορούν να μετακινούν ελεύθερα στην ε, Γερμανία ή την ε, Ολλανδία για να δουλέψουν και υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Λοιπόν, η Γερμανία έχει συγκρατήσει το κόστος της συμπεριλαμβανομένων και των φόρων και των μισθών. Ως εκ τούτου πέτυχε να κερδίσει ανταγωνιστικότητα και το έπραξε ότι γνωρίζαμε ότι η αύξηση του κόσμου εργασίας θα πρέπει να ε, πηγαίνει χέρι-χέρι με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν διαφορά σε αυτά τα επίπεδα και τότε αυτό δημιουργεί προβλήματα σε μια ζώνη που δεν είναι πολιτικά ολοκληρωμένη και από τις δύο πλευρές θα ειδικά όταν μιλάμε για συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν, του Συμβουλίου Υπουργών και από οικονομολόγους εμπειρογνώμονες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να ε, υποστούν κάποιο κόστος προσαρμογής, να πληρώσουν κάποιο κόστος προσαρμογής. Φυσικά συμφωνώ και αυτό είναι το τελευταίο σημείο μου ότι το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να πέσει στις ελληματικές χώρες. Αλλά οι χώρες που έχουν πλεονάσμα έχουν, φέρουν κάποια ευθύνη και η προσπάθεια αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, βελτίωσης μάλλον, είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας αποσχολεί όλους. Ωραία, κύριε Πιζάνη, Φέρη Σε πολλά έχετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αν και καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να υποκαταστήσω τους εκπροσώπους των θερμικών οργάνων που ακούστηκαν πριν από εμένα. Να πω καταρχάς ότι υπάρχει κάποια μικρή παρανόηση. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι πρέπει να ανησυχούμε. Τα επίπεδα των ελλημάτων όπως διαπιστώσαμε μετά την έναρξη της κρίσης ήταν λόγος ανησυχίας. Αυτό που λέω είναι ότι για το δημόσιο έλλειμμα έχουμε κάποια όρια για το τι θεωρούμε αποδεκτό ή όχι. Αλλά όταν μιλάμε για το ισοζύγιο, ποτέ δεν γνωρίζουμε τι είναι καλό ή κακό όσον αφορά τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα. Και βεβαίως πρόκειται και για κάτι που είναι βιώσιμο, γιατί μπορεί να επιτρέψει την αύξηση των εσόδων στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά όμως, αν το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου μπορεί να οφείλεται σε αύξηση της κατανάλωσης ή των κατασκευών, τότε μπορεί κάποια στιγμή αυτή η φούσκα να καταρρεύσει και να έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα κάποιες χώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να βασιζόμαστε στην αυτοδιόρθωση των προβλημάτων. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι οι δυνατότητες αυτοδιόρθωσης ήταν πολύ αδύναμες οι αγορές μας δεν ήταν αρκετά ενοποιημένες προκειμένου να μπορέσουν να αντιδράσουν άμεσα. Και αυτό που διαπιστώσαμε επίσης είναι ότι οι φούσκες μπορεί να αναπτύσσονται για πολύ καιρό, να αναπτύσσεται η οικονομία όπως γινόταν στην Ισπανία και την Ιρλανδία και μετά να καταλήγουμε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση από την οποία πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο για να προσαρμοστούμε. Τώρα, το ποιος πρέπει να προσαρμοστεί. Ας δούμε καταρχάς τους αριθμούς. Μας είπατε ότι δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί στην Πορτογαλία από την εισαγωγή του ευρώ. Εγώ όμως αυτό που βλέπω στις στατιστικές είναι ότι η ονομαστική μισθή στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 43% και κατά 25% στη Γερμανία. Αυτή η αύξηση οδήγησε και σε αύξηση τιμών. Ίσως λοιπόν δεν είχαμε αύξηση της αγοραστικής δύναμης, αλλά οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν και ενδεχομένως είναι υπερβολικά υψηλοί στη χώρα σας και κάποιες άλλες χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε την τιμή παντού και ταυτόχρονα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν καλή λύση, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο σε πολύ μικρές κλειστές οικονομίες όπου έχουμε συνειδητοποιημένους πολίτες που είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν κάτι τέτοιο γιατί θα βλέπουν αμέσως τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία. Αυτό όμως δεν ισχύει για την Ισπανία που δεν είναι τόσο ανοιχτή οικονομία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλή λύση για την Ισπανία. Στις ε, χώρες λοιπόν που δεν έχουν τόσο ανοιχτή οικονομία θα χρειαστεί μία σταδιακή ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας όπως είχε γίνει στην Γερμανία ή στη Γαλλία τη δεκαετία του 80. Τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε την ανάκαμψη. Η αύξηση των μισθών στη Γερμανία θα μπορούσε να βοηθήσει τους εταίρους ενώ το πάγωμα των μισθών σε ορισμένους τομείς δεν βοηθάει. Οι μισθοί πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την παραγωγικότητα και με τους στόχους για τον πληθωρισμό. Αυτό θα βοηθούσε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως αυτό δεν είναι εργαλείο πολιτικής. Δεν μπορεί να αποφασιστεί σε κυβερνητικό επίπεδο. Ειδικά σε χώρες όπου δεν υπάρχει συγκεντρωτική απόφαση για συλλογικές συμβάσεις όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Κάποια σχόλια για τη στρατηγική του για το 2020, επειδή πολλοί το ανέφεραν. Υπήρξε ένα ερώτημα για το τι σχέση έχει αυτή η στρατηγική με τη σημερινή κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοιου είδου στρατηγική τώρα. Γιατί πριν την κρίση θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε πορεία ύφεση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η απασχόληση αυξάνεται, έχουμε μικρή ανάπτυξη αλλά ανάπτυξη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα επερχόμενα χρόνια. Τώρα έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε που οφείλεται στα δημοσιονομικά προβλήματα και φοβούμαστε τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου όπου θα έχουμε χαμηλή ανάπτυξη, όπου τα δημοσιονομικά προβλήματα θα παραμένουν παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των ελλημάτων και τέτοιου είδους παραδείγματα έχουμε στην ιστορία με φαύλους κύκλους στασιμότητας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν με τη στρατηγική. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα σε επίπεδο διακυβέρνησης. Αναφερθήκαμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους νέους που βεβαίως πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική. Τα εργαλεία όμως ποια είναι. Οι κυρώσεις. Σας είπα ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για κυρώσεις. Μπορούμε όμως να συγκρίνουμε αποθάσεις και να αυτές τις συγκρίσεις να τις κάνουμε πιο γνωστές και πιο διαφανείς, να τις γνωρίζουν οι πολίτες, να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση των κυβερνήσεών τους. Αυτό είναι κάτι που δεν είχε περάσει στη στρατηγική της Λισαβόνας γιατί κανείς δεν ήθελε αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρόοδο εδώ και να έχουμε πίνακες συγκριτικούς, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Και αυτό θα βοηθούσε και τη δημοκρατικό διάλογο. Γιατί αν επιλέξουμε τους κατάλληλους δείκτες θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την πορεία μας σε σχέση με αυτή των γειτόνων μας. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν προκλήσεις. Θα ήθελα όμως να καταλήξω με μια αισιόδοξη νότα. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ κακά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Δεν ήταν προετοιμασμένη για την κρίση του τραπεζικού συστήματος. Όλοι γνωρίζαμε ότι το σύστημα ήταν μεταβατικό μεταξύ της κατάστασης όπου όλη την ευθύνη θα την έφερε το εθνικό επίπεδο και της ε, νέας κατάστασης όπου θα είχαμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση δεν είχαμε βέλτιστη δημοσιονομική σταθερότητα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε κίνητρα και σε εθνικό επίπεδο προϋπολογισμού. Βρισκόμασταν σε δύσκολη θέση όταν άρχισε να αντιστρέφεται η πορεία των ροών κεφαλαίου. όταν σταμάτησε η μαζική ζωή κεφαλαίων σε ορισμένα κράτη-μέλη παρόλα αυτά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όχι τέλεια, αλλά καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε λοιπόν να εξάγουμε πολλά διδάγματα, γιατί σε μια δύσκολη κατάσταση βρήκαμε λύσεις. Για παράδειγμα, στο χρήση των τραπεζών. Επίση υπήρξε η λύση με τα πακέτα κινήτρων. Υπήρξε η πρωτοβουλία της Βιέννης. Μπορούμε λοιπόν να εξάγουμε μαθήματα και να μάθουμε από τα λάθη μας, να μάθουμε από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που διαπιστώσαμε στις πολιτικές μας και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα προσεγγίζουμε την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, το πέρας της. Δεν θα καταλήξω σε συμπεράσματα σε σχέση με το ποιες θα ήταν οι προθέσεις ε, των συμπροευρωμένων. Εδώ έχω όμως κάποιες ε, σημειώσεις για κύρια στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν. Συνολικά υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι χρειάζεται περισσότερος συντονισμός, συντονισμός ε, της οικονομικής πολιτικής στο οικονομικό πολιτικό επίπεδο και υπάρχουν ευκαιρίες να γίνει αυτό τώρα, μια και έχει επικυρωθεί η συνθήκη της Σαβώνας. Είναι ενδιαφέρον να ακούσει κανείς αυτό που είπε όλοι Ρέν, ότι χάσαμε 20 χρόνια εξυγίανσης τα τελευταία δύο χρόνια των δημοσιονομικών μας και πρέπει τώρα να, να, καλύψουμε αυτό το κενό. Αυτό. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Ο κύριος Στάκ είπε ότι άνηση θα είναι λέει ανάπτυξη και τομεακά άνηση και αναχώρα άνηση και τα λοιπά. Και γι' αυτό πολύ ανέφεραν επίσης την ανάγκη να έχουμε ένα είδος οροσίμων ή μετρήσεων καθοδόν προς το 2020 και πιο σημαντικό ακόμα σε σχέση με τις ανισότητες στην ανάπτυξη να αντιμετωπιστούν. Αναφέρθηκε ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και σίγουρα θα ακούσουμε κάτι παραπάνω απόψε όσον αφορά τον Μάριο Μόντι, κύριο μιλητή για αυτά τα θέματα. Υπήρξε αναφορά στην ανάγκη της μεταρρύθμισης του οικονομικού προτύπου μας με, καλύτερα μέσα, καλύτερους μηχανισμούς διασφαλίζοντας ότι θα είναι συμβατά και θα συνάδουν όλα αυτά και να μην εξαρτώμαστε μόνο στην ε, ισορροπία των ε, ε, δημοσιονομικών και της φορολογίας. Το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει ένα οικολογικό όριο όσον αφορά τις στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν και να εκτελεστούν και μην ξεχνάμε φυσικά ότι οι σε επιχειρήσεις, η ΜΜΕ είναι ο κινητήρας, η κινητήρια δύναμη για μας και για αλλού παγκόσμια. Και για μια επιπλέον θέση απασχόλησης σε κάθε μικροεταιρεία, αν δημιουργούσαμε μια τέτοια άνα θα υπαρκούσε να επιληθεί το πρόβλημα απασχόλησης. Αυτά πρέπει να λυθούν υπόψη στην πορεία προς τα εμπρός. Ακόμα και οι μικρότεροι και οι έσχατοι μπορούν να βοηθήσουν για να διασωθούμε όλοι. Αυτά ήτανε ε, λυπούμε για την αποχώρηση κάποιων ομιλητών. Θα αναλυφθούν μέτρα και διαβήματα ώστε να μην συμβεί αυτό, να μην επαναληφθεί ακόμα και αύριο. Έχω υπόψη μου κυρώσει ε, εντό εισαγωγικών για αυτού που αποχώρησαν ε, ε, σήμερα. Έχουμε κάποια πράγματα υπόψη. Τώρα, για τους μηχανισμούς, για το τι θα γίνει απόψε. Λοιπόν, όσοι από εσά θα έρθετε για το δείπνο, να σας υπενθυμίσω, θα γίνει στο ισόγειο, θα παρασχεθεί, θα παρατεθεί, στο ισόγειο, επίπεδο 0 δηλαδή, ισόγειο, για το, στο εστιατόριο των μελών. Από τις 6.30 και περαιτέρω θα σερβίρονται ποτά. Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής, Γέρζι Μπούζεκ, θα σας καλωσορίσει στις 7 η ώρα. Προτού ο κύριος Μάριο Μόντι, φιλοξενούμενος αγορητής, προσέχει να παρέμβει. Δεν είναι καλή ιδέα να εγκαταλείψετε το κτίριο πριν από το δείπνο, γιατί θα υπήρχε ίσως δυσκολία να επανέλθετε. Και καθώς έχετε κάποιες ευφυείς ρυθμίσεις, ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορεί καλύτερα να λειτουργήσει κανείς. Θα επανέλθουμε αύριο εδώ το πρωί στις 9.00. 09.00 και θα ε, θα πρέπει έτσι να προσδέσουμε τους κύριους αγορητές για να μην εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ευχαριστώ.